Καλημέρα σα, συνάδελφοι. Θα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μήπω αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. Τώρα μερικέ αλλαγέ. Το σημείο 3 ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής με τον κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο αναβάλλεται. Θα το συζητήσω με τους συντονιστές γιατί τόσο καθυστερημένα έγινε αυτή η αλλαγή. Δεν είναι σωστό αυτό. Θα κάνουμε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων για τον δομημένο διάλογο μετά από τη συνεδρίασή μας και το θέμα του κυρίου Αβραμοπούλου θα τεθεί στους συντονιστάς. Θα έρθει άλλη φορά βέβαια, αλλά πάντως εμείς θα το συζητήσουμε. Έπειτα, για το σημείο 8 του σχέδιου τροπολογία 5 στο Γενικό Προπολογισμό 2015 ανταπόκριση στι μεταναστευτικέ ροέ και πιέσει. Αυτό θα γίνει 10 και 4 αντί για. Point 10 on the petition on Spanish security law. This is going to be postponed. And also, if I, colleagues, if I have your attention, point 6 on EU PNR uh, will be postponed. Our rapporteur, again, at fairly late notice, um, could not be here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 και αμέσως μετά την ψηφοφορία στις 3 μάλλον και παρακαλώ στις 3 να έχετε και τις κάρτες σας τις κάρτες Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ακόμα και αν θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχω ενοχληθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να συναντήσουμε τον Φράσ Τίμερμανς και μας ακύρωσε τελευταία στιγμή. Σήμερα θα είχαμε δομημένο διάλογο με τον κύριο Αβραμόπουλο που πάλι αναβλήθηκε. Δεν είναι εθελοντικό και άμα θέλουν έρχονται οι επιτροποί. είναι στην διοργανική συμφωνία και πρέπει να ολοκληρωθεί νομίζω αυτή την εβδομάδα και αναρωτιέμαι ποια δικαιολογία έχουν. Γιατί δεν γίνονται αυτοί οι διάλογοι και θα με ενδιέφερε επίσης γιατί το σημείο του Ισπανικού νόμου ασφαλείας δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Πρέπει κάποτε και η Κομισιόν νομίζω να είναι σε θέση να τοποθετηθεί από αυτό. Thank you for that. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο για την απουσία ε, των ε, δύο επιτρόπων για τον ε, δομημένο διάλογο. Αλλιώς να απαντήσω σε αυτά. Ναι, πρώτα απ' όλα έχετε δίκιο για το θέμα της απουσίας του κυρίου Αβραμόπουλου από τον δομημένο, του, από τον δομημένο διάλογο. Δεν είναι μια κοινωνική επίσκεψη είναι μέρος του δομημένου διαλόγου που πρέπει όλες οι επιτροπές να έχουν στο πλαίσιο της διαδικασίας της διάσκεψης των Πρόεδρων που πολύ σωστά είπατε έχει προθεσμίες. Μας ενημέρωσε τελευταία στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Αβραμόπουλος πως για προσωπικούς λόγους δεν ε, μπορούσε να έρθει σήμερα και προφανώς ε, τους είπα πως είναι πολύ προβληματικό αυτό και θα έχουμε μόνο την κυρία Γιώργα. Θα το θέσω στους συντονιστές, όπως είπα, για να δούμε τι θα κάνουμε παραπέρα. Γιατί είναι σοβαρό ζήτημα δεν έχουμε πλέον δομημένο διάλογο. Προφανώς λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει και το ζήτημα του κυρίου Τίμερμανς και του τι θα μας πει. Και θα το θέσω στους συντονιστές, αλλά και εσείς καλά τα είπατε. Θα το θέσω λοιπόν στους επιτρόπους και θα σας ενημερώσω. Είναι πράγματι σοβαρό. Για το θέμα του Ισπανικού νόμου η Κομισιόν δεν ήταν διαθέσιμη, γι' αυτό αναβλήθηκε. Δικαίως όμως ε, είστε εκνευρισμένοι. Εγκρίνεται η μερίσχη διάταξη λοιπόν. Σόφι Νετφέλτ. Την ίδια ερώτηση θα έκανα κι εγώ. η Κομισιόν ε, δεν ε, ήταν διαθέσιμη. Μα τι σημαίνει αυτό. Είναι σοβαρό θέμα. Γιατί μη διαθέσιμη σημαίνει ότι μου είπαν ότι δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό σημαίνει. Ε, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή. Δεν θέλω να να μην είμαι ειλικρινής. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα είναι πάντως στη διάθεσή μας στην επόμενη συνεδρίαση. Και ζητώ συγγνώμη. Συνάδελφοι, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Ωραία, περνάμε άρα στο σημείο 2 Το ανακοινώσεων του Προέδρου. ερμηνεία σε πολλές ε, γλώσσες ε, δανέζικα, λετωνικά, κροατικά και ε, γοεδελικά δεν υπάρχουν το πρωί και το απόγευμα λοιπόν για τις αποφάσεις των συντονιστών αποφασίσαμε να υποβάλουμε Parliament resolution of the 11th of February on the US Senate report on the Δεύτερον, χρήση βασανιστήριων από την CIA και η συνέχεια στη σχετική έκθεση. Αποφασίσαμε να συσταθεί μια άτυπη ομάδα εργασίας με ένα μέλος από κάθε πολιτική ομάδα υπό την Προεδρία του Πρόεδρου για να προετοιμάσουμε την ακρόαση και την αποστολή. Καθώς ε, βεβαίως ε, θα πρέπει εδώ πέρα να εμπλακεί και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα μέλος ε, της ε, ΑΦΕΤ ε, και ειδικά της Επιτροπής ΑΦΕΤ, της Επιτροπής ΔΡΟΑ μπορεί να συμμετάσχει. Λοιπόν, Παράγραφος 20 του ψηφίσματος 11 Μαρτίου 2015 για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο αποφασίσαμε να συντάξουμε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας υπομορφή έκθεσης ε, εφαρμογής του θέματος ε, αυτού κατόπιν. η επόμενη συνεδριάση 26 Μαΐου μισή μέρα 1η Ιουνίου μισή μέρα, 25 Ιουνίου, ολόκληρη ημέρα. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε και άλλες συνεδριάσεις στις 26 Μαΐου και στις 25 Ιουνίου. Πρόσκληση για να οριστεί μέρος της Επιτροπής μας, το οποίο θα πάει στην Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Ένωση. Αποφασίσαμε να ορίσουμε τον κύριο Μπόνι. Εγκρίνεται λοιπόν τις συστάσεις αυτές των συντονιστών. Ωραία, καμία αντίρρηση. Εγκρίνονται λοιπόν αυτά. Τέλος και πάλι να σας υπενθυμίσω πως έχουμε μία ψηφοφορία στις 3 η ώρα. Φέρτε λοιπόν τις κάρτες σας. Έχουμε λοιπόν δύο σημαντικά θέματα. Ξεκινάμε με το σημείο 3. Ο διαρθρωμένος διάλογος και τουλάχιστον μία επιτροπός ήρθε Συγχαρητήρια. Ε, ξέρετε τώρα πως ε, είμαστε εδώ πέρα. Και πετάξατε σήμερα το πρωί. Μπράβο, μπράβο. Όταν λοιπόν τους ξαναδείτε τους άλλους εκεί πέρα, πείτε στον κύριο Αβραμόπουλο και στον κύριο Τίμερμανς ότι η διάσκεψη των Προέδρων απαιτεί να τηρούν τα ραντεβού. Μέλος, μέλος με συγχωρείτε, του διαρθρωμένου διαλόγου είναι έγκριση του προγράμματος ε, και εφαρμογή του προγράμματος 2015, προτεραιότητες για το 2016 και βεβαίως να ενημερωθούμε για το τι θα γίνει στο μέλλον. για το πρόγραμμα εργασίας. Οπότε προφανώς το δούμε το δικό σας χαρτοφυλάκιο, θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και νέες πρωτοβουλίες, ε, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που είμαστε με τα δικονομικά δικαιώματα και τα λοιπά. Και ξέρω βέβαια πως σας απασχολούν αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και έχετε 10 ε, λεπτά για να κάνετε μια εισαγωγή ειδικά για το άμεσο μέλλον και μετά θα ακούσουμε τους συντονιστές και τους βουλευτές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε λοιπόν, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράες, αξιόδημοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Κέρδισα το βραβείο που κατάφερα να έρθω εδώ. Ελπίζω όμως ότι στο τέλος της μέρας δεν θα μου το έχετε πάρει πίσω. Και να σας απαντήσω στις τυχόν ερωτήσεις που θα αντιστοιχούσαν και στο συνάδελφο Αβραμόπουλο γιατί τα χαρτοφυλάκια μας είναι πολύ σχετικά ασφάλεια κλπ. Έχει βέβαια και κάποια συγκεκριμένα θέματα στο χαρτοφυλάκιό του οπότε βέβαια σε κάποια άλλη ευκαιρία θα μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για ό,τι αφορά εκείνον. Πάντως σήμερα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε Είχαμε πει τότε που άρχισε η εντολή μου ότι θα ήθελα να έχω συνεχή επικοινωνία μαζί σας. Σε τακτά διαστήματα. Που είναι για μένα μια ευκαιρία να σας ενημερώνω. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας για το 2016. Οπότε και έτσι θα μου πείτε και εσείς τις προτάσεις σας για αυτό το πρόγραμμα. Όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη, φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποιες προτάσεις για το τι θα κάνουμε το 2016. Η ομιλία μου θα επικεντρωθεί περισσότερο στο 2015. Άρα την τρέχουσα νομοπαρασκευαστική διαδικασία και θεματολόγιο. Να δούμε τι θα γίνει με την προστασία των δεδομένων και να δούμε για αυτή τη μεταρρύθμιση του δικαίου της προστασίας των δεδομένων τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε σε σχέση με τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Επίσης, θα μας απασχολήσουν η οδηγία, η διαβρύνση της απάτης, τα δικονομικά θέματα, η Eurojust, με κάποιες νέες πρωτοβουλίες σχετικά με το θεματολόγιο της ασφαλείας, επίσης του Μητρώου και της ριζοσπαστικοποίησης της φυλακής. Το έκρις τώρα, το σύστημα αυτό ε, στις 28 Απριλίου εγκρίναμε το θεματολόγιο για την ασφάλεια που γνωρίζετε και θέλουμε αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών. Πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις τωρινές απειλές στην ασφάλεια. Σήμερα έχουμε 26 κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα εκρή που αφορά τα ποινικά μητρώα. Αφορά προηγούμενες καταδίκες για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάποιους πάντω δεν είναι τόσο αποτελεσματικό το σύστημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εξολογεί το πώ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και ταυτόχρονα να λάβει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προσοχή των δεδομένων. Και μέσα στι επόμενε εβδομάδε πρόκειται να διερευνήσουμε ποιο είναι ο πιο δόκιμο τρόπο να το κάνουμε αυτό. Θα επιταχύνουμε το έργο το οποίο ήδη αρχίσει, ούτω ώστε το έκρης για πολίτες χωρών εκτός ένωσης θα βελτιωθεί και πώς το έκρης θα εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά. Δύο λόγια τώρα όσον αφορά την οδηγία του τη της απάτης. Χαιρετίζουμε την ε, πρόοδο των συνομοθετών όσον αφορά αυτή την ε, οδηγία αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένα συμβασμό για δύο. την πρώτα-πρώτα το να καλύψουμε τον ΦΠΑ ε, και κάποιες ε, κυρώσεις καθώς επίσης και τις προθεσμίες παραγραφής για κάποια δικήματα για να δούμε πώς θα φραγίσουμε το, το νομοθετικό πλαίσιο να προσταθούμε τα συμφέροντα της κοινότητας και να μην υποχωρήσουμε πουθενά στον αφορά την προστασία αυτή βάσει της νομοθεσίας. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Δηλαδή θα έχουμε χειρότερη ρύθμιση από τη ε, Συμφωνία του 1995 αν κολλήσουμε αυτό που λέει το Συμβούλιο για τον ΦΠΑ. Οπότε θα πρέπει τώρα αυτή η οδηγία να είναι κάτι το οποίο να συνάδει προς τις δικές μας ε, φιλοδοξίες. Επίσης, η, αυτή η οδηγία ε, σχετίζεται με την υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Έχουμε την κυρία Μαγκοβέ, έχουμε τους άλλους και οι οποίοι για αυτό το δύσκολο θέμα έχουν κάνει πάρα πολλά. Και στις 29 Τετάρτου εγκρίθηκε η ενδιάμεση έκθεση όσον αφορά ε, την γνώμη σας για την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Και εσείς όπως και εμείς θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια ανεξάρτητη υπηρεσία και να είναι και αποτελεσματική. Και θέλουμε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή υπηρεσία, να έχει διασυνοριακές ε, ε, αρμοδιότητες έρευνας και αυτό για όλο το ε, αδιέρετο και όλο το προσωπικό και τους αντισαγγελείς. Οπότε θέλουμε να δούμε τι έχει να πει το ΔΕΚ, γιατί το ΔΕΚ είναι ο αυθεντικός ερμηνευτής του κοινωτικού δικαίου. Θα πρέπει στους αμέσους μήνες να μπορέσουμε να εργαστούμε εντατικά πάνω στο κείμενο που έχουμε και να δούμε τι προστιθέμενη αξία θα προκύψει και εμείς δεν θα αφιστούμε προσπαθειών ώστε η εισαγγελία να έχει συγκροτηθεί μέχρι το 2016 όπως προβλέπει το πρόγραμμα του Πρόεδρου Γιούγκερ και γι' αυτό και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την μεταρρύθμιση της Eurojust και την ολοκλήρωση των οικονομικών δικαιωμάτων. Θα συνεργαστούμε για όλα αυτά πολύ στενά με τους συζητητές. Δύο λόγια τώρα για το σημαντικό πρόβλημα το σημερινό, δηλαδή την ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Στα πλαίσια θεματολογία την ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδώσει μεγάλη σημασία στο πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση που ε, συνήθως γίνεται μέσω του διαδικτύου και στις φυλακές. Οπότε τα θέματα τη κράτη και φυλάκιση είναι θέματα εθνικού δικαίου. Αλλά η αντιμετώπιση τη ε, στρατολόγηση ε, τρομοκρατών και τη βαστικοποίηση ε, στα συγχρονιστικά κέντρα είναι κάτι το οποίο απαιτεί ευρωπαϊκέ προσπάθειε. Για να μπορέσουμε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, έχουμε μια ομάδα εργασία για τι φυλακέ, για την αναστολή των ποινών και θα κάνουμε και στι 19 και 20 δεκάτου μια, μια, μια διάσκεψη ε, υπό την αιγύδα της Προεδρίας του Συμβουλίου. Θα έχουμε, θέλουμε ανταλλαγή απόψεων, να δούμε τι θα γίνει με ριζοσπαστικοποίηση, θα γίνει με τις ε, ιδέες χρήσης της βίας, κάτι το οποίο εξαπλώνεται στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ με το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την πρόληψη ε, της ζωστικοποίησεις και επίσης να εκπαιδεύσουμε και πρόσωπο που θα ασχοληθεί με αυτό και επίσης θέλω να είναι το ευρύτερο πλαίσιο του θέματος της ε, κράτησης στα πλαίσια της εκθεσιδίας πρωτοβουλίας. Τώρα για να δούμε τι γίνεται με τη μεταρρύθμιση των ε, νόμων, των διατάξεων για την των δεδομένων. Αυτό είναι η ψήστη προτεραιότητα για φέτος. Και με χαρά μου πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την πρωτοπόρα γνώμη σας για αυτό το θέμα, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και στα πλαίσια του Συμβουλίου, όπου πετύχαμε αρκετή πρόοδο στις τελευταίες συναντήσεις, στα τελευταία συμβούλια, οπότε πιστεύω ότι στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης του Ιουνίου πρόκειται να πετύχουμε μια γενική προσέγγιση και αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά θα μπορέσουμε να αρχίσουμε ε, τους κοινωνικούς διαλόγους, ούτω ώστε με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει να ολοκληρώσουμε την μεταρρύθμιση για φέτος και η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για λιγοστή των δεδομένων τώρα γνωρίζει καινούργια όθηση γιατί είχαμε ε, το θυματολόγιο για την ενιαία ψηφιακή αγορά που δίθηκε τώρα πρόσφατα και έτσι με αυτή την αγορά μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και περιμένω πώς και πώς να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για την επόμενη φάση, τη φάση του τριγωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων. Επίσης, προσθέτω ότι ακόμα έχω ελπίδες ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις επαφές με τις ΥΠΑ για τη Συμφωνία Ομπρέλα και για τον ασφαλή λιμένα. Υπάρχουν κάποια θέματα που ακόμη εκκρεμούν, ε, είναι σκληρές διαπραγματεύσεις αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε κάτι να προκύψει. Πρόεδρε. Έχουμε την αρχική διάταξη στο θεματολόγιο της ασφάλειας και τι λέει ότι θα πρέπει σε αυτή την περιοχή ελευθερίας, δικαιοσύνης και ε, δημοκρατίας και ασφάλειας θα πρέπει να κάνει η Επιτροπή ότι μπορεί για να τους παράγει την ασφάλεια. Οπότε θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι να ξέρουν ότι όπου μετακινούνται στην Ευρώπη η ασφάλειά τους και η ελευθερία τους είναι προστατευμένες. Ακριβώς όπως ε, προβλέπουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και πάλι σας ευχαριστώ για την στήριξή σας σε όλα αυτά τα θέματα και περιμένω την ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε τον χρόνο και ήρθατε εδώ. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας γιατί και ξέρω ότι τα μέλη μας θα έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε με τις ερωτήσεις των συντονιστών. Και να σας πω πως χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω για να μπούμε σε λεπτομέρειες και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ε, προτεραιότητες λοιπόν για το 2016 και εφαρμογή του προγράμματος του 2015. Θα αρχίσουμε με την κυρία Χολμάιρ, συντονίστρια του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το 2016 και τι θα γίνει το 2016 σχετικά με τους ε, τριμερείς ε, διαλόγους οι οποίοι διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Έπειτα, Eurojust. Θα ήθελα να πω πως καλωσορίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη στον ε, τομέα της δικαστικής συνεργασίας και στηρίζει και προσωπικά την Eurojust. Πιστεύω πως είναι πολύ αναγκαία η επίσπευση των ε, νομικών διαδικασιών, των δικαστικών ε, διαδικασιών και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν ε, αναγκαίο το συντονιστικό έργο της Eurojust. Από τη μία η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από την άλλη όμως είναι εξίσου σημαντική και η επάνδρωση της Eurojust. Έπειτα, όσον αφορά το ζήτημα της απάτης, ζητούμε το θέμα της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πιστεύω πως δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πιστεύω πως τα κράτη-μέλη καθυστερούν. Ωστόσο θα με ενδιαφέρει να μάθω εσείς τι άποψη έχετε για την προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από νομική άποψη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις οικονομικών ε, ζημιών, για παράδειγμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Πρόκειται για ζημιές ε, δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα, μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα προγράμματα στο ΕΦΣΙ για παράδειγμα. Ε, τώρα, μία άλλη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες ιδέες για το πώς θα διεξαχθούν οι διαδικασίες ελέγχου με τις Ηνωμένε Πολιτείες μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη Διεθνική Συμφωνία. Και έπειτα μπορεί να υπάρχει η λέξη έλεγχος στην συμφωνία, όμως τι σημαίνει πραγματικά αυτός ο έλεγχος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συντονίστρια από τους Σοσιαλδημοκράτες, κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ περισσότερο στο πρόγραμμα εργασίας του 2016 και συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς. Καταρχάς, θεμελιώδη δικαιώματα. Και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Δεδομένων των συνεχιζόμενων δυσκολιών στην ε, ένταξη των, ιδιαίτερα των ε, Ρωμά στην Ευρώπη και δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασία του 2016 συγκεκριμένα στοιχεία ε, που θα αναφέρονται σε στρατηγικέ ένταξει των Ρωμά και εάν ναι, ποια στοιχεία είναι αυτά. Επίση, η κυρία Επίτροπο ε, αναλαμβάνει δέσμευση για δημιουργία στρατηγική για του ΕΛΟΑΔ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αρκετές φορές να γίνει κάτι τέτοιο. Θα παρουσιάσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασίας μια στρατηγική για τους ε, ΛΟΑΔ και εάν όχι γιατί. Έπειτα, ποινικό δίκαιο. Στην έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ιανουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση για να επιλύσει τα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή ε, της απόφασης πλαίσιο του 2015 ε, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Υπάρχει κάποια πρόταση για ένα οριζόντιο όργανο το οποίο θα ξεπεράσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει και θα ε, υπάρξουν επίσης μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης το ποινικό δίκαιο ή υπάρχει κάποια πρόταση για αναθεώρηση της απόφασης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπεριλάβει μια τέτοια πρόταση στο πρόγραμμα εργασίας της. Και τρίτον, η προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την προστασία προσωπικών δεδομένων ε, ε, υπό το πρόγραμμα του Safe Haven. Ε, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθήκων σκοπεύει να το διορθώσει αυτό. Και το πρόγραμμα Safe Haven είναι συμβατό με τις συνθήκες. Έπειτα, σχετικά με την μεταρρύθμιση της αρχής στα προσωπικά δεδομένα, μας ε, αναφέρεται πως πρόκειται να διεξαχθούν διαθρωμένοι διάλογοι αυτό το καλοκαίρι. Θα συμπεριλάβουν και τον κανονισμό ή ε, μόνο την οδηγία, διότι εμείς ζητήσαμε να γίνει συζήτηση για όλο το πακέτο των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στίβενς για την ομάδα ECR. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι προηγούμενοι. Αλλά βλέπω πως έχετε πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα της μη διακριτικής μεταχείρισης ατόμων με βάση το φύλλο, την αναπηρία κτλ. Επίσης η προστασία των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό ναι. θέμα και πρέπει να αναθεωρηθεί, να εξυγχρονιστεί. Και τρίτον, έχουμε τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ για την προστασία των δεδομένων και των ασφαλή λιμένα. Και τέλος, θα γίνει η συζήτηση για την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα επανέλθω σε αυτό. Σημείωσα επίσης πως ε, υπάρχουν και άλλες ακόμα προτάσεις επιτάπητος όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Η Κομισιόν ε, πρέπει να εστιαστεί σε ίσες ευκαιρίες για όλους. Άνδρες, γυναίκες, ε, ΛΟΑΔΑ, ε, ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και βεβαίως ε, άτομα με αναπηρίες. Νομίζω λοιπόν πως για όλα αυτά δεν έχουμε κάνει κάποια πολύ σοβαρή γενική συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την άλλη κυρία Ινετφέλτ Σόφη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Mm. Καλωσορίσατε κυρία Επίτροπέ μου. Χαίρομαι για την παρουσία σας. Καταρχάς, ο Επίτροπος Τίμερμανς ανακοίνωσε ότι στη νέα διαθεσμική συμφωνία θα συμπεριλάβει μια ρήτρα που θα λέει ότι αν το Κοινοβούλιο ζητήσει νέα προγράμματα ή νομοθετικές πρωτοβουλίες, τότε η Κομισιόν είτε θα δεχτεί αυτή την πρόταση είτε θα πρέπει να δικαιολογήσει γιατί δεν τη δέχεται. Καλό είναι αυτό, διότι η Κομισιόν έχει αυτή την υποχρέωση για τις πρωτοβουλίες των πολιτών και την ίδια υποχρέωση θα έπρεπε να έχει και ως προς τις αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρία θέματα θέλω να θίξω, δύο τα είπαν οι προηγούμενοι. Επανειλημμένως έχουμε ζητήσει να ακυρωθεί το λεγόμενο safe harbor, ασφαλής λιμίν. Δεύτερον, μία στρατηγική πρόγραμμα για τους LGBT και τρίτον, την αποτίμηση, την αξιολόγηση των προγραμμάτων καταπολέμησης της τραμακρατίας. Ελπίζω να τα συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα εργασιών. Έπειτα. Μία από τις προτεραιότητές σας είναι η οριζόντια οδηγία ίσης μεταχείρισης. Ξέρω ότι είναι δικαιοδοσία των χωρών μελών, αλλά ανακοινώσατε όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας ότι θα πιέζατε πολύ για να εγκριθεί αυτό που είναι τα πράγματα λοιπόν και τέλος, τέλος Δύο θέματα που θα ήθελα η Κομισιό να συμπεριλάβει επίσης στο πρόγραμμα εργασιών της είναι το ένα κάποιο πλαίσιο ή μηχανισμό για ετήσια αξιολόγηση όλα τα κράτη-μέλη της κατάστασης της δημοκρατικής διακυβέρνησης και του σεβασμού ημί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν λέω να συζητάμε συνεχώς τις ίδιες χώρες, αλλά ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όλες οι πολιτικές ομάδες λίγο πολύ το έχουν ζητήσει. Ένα μηχανισμό δηλαδή αξιολόγηση στην κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Και το δεύτερο, ξέρετε ότι σε μερικές χώρες μέλη υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται Child Alert για τις εξαφανίσεις παιδών είναι θελοντικό πρόγραμμα αλλά θα ωφελούνταν πολύ από ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαστικών αρχών και αστυνομίας και η Κομισιόν ήδη χρόνια πριν ανακοίνωσε ότι θα μελετούσε την περίπτωση να αναλυθεί μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία και ελπίζω να το συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα Σας Ευχαριστώ. πολύ. Ο κύριος Χρυσόγονος για την ΚΟΕ. Thank Chairman. Uh, welcome, Commissioner. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Στο οικιά σα προβλέπετε το να ε, ολοκληρώσετε τη σύναψη της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά την προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οπότε, θα σε ρωτώ πρώτα πρώτα. Πώς προτίθεστε να απεμπλέξετε την κατάσταση που τώρα έχει εμπλακεί μετά την, τελευ... πρόσφατη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου όσον αφορά την ε, προσχώρηση. Και σε σχέση με αυτό σας υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε μόνο τα δικαιώματα υπεράσπισης που προβλέπονται στον χάρτη των δικαιωμάτων. Έχουμε επίσης και τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από τον χάρτη των δικαιωμάτων. Άρα δεν θα ήταν ε, καλή ιδέα να προλιάνουμε το έδαφος για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον χάρτη των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο τώρα. Αφορά τη διαφθορά. Έχουμε πρόσφατες δημοσιεύσεις της ε, διεθνούς διαφάνειας και λέει ότι όχι μόνο τα μέλη αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλά θα πρέπει ακόμα να γίνουν για τη διαφθορά και σε σχέση με την παράτυπη χρήση κοινωνικών πόρων. Δεν έχει ακόμα αναγκαστεί τίποτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την διαφθορά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε, πότε προβλέπετε να δημοσιοποιήσετε μια έκθεση για αυτό το θέμα. Πότε θα θίξετε όλες αυτές τις πλευρές του προβλήματος. Τρίτη και τελευταία ερώτηση τώρα. Από ό,τι διαπιστώνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σταματήσει να είναι πρωτοπόρα στον τομέα της ισότητα. Πώς θα διστρέψει αυτή την τάση το 2015, αλλά και μέσα από το πρόγραμμα εργασιών και το 2016 και ιδίω με ανάπτυξη πρωτοβουλίου. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Ολμπρικ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ. Έχω μόνο μια ερώτηση όσον αφορά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πώς θα υλοποιηθεί ο χάρτης για τους ΛΟΑΔ. Έχετε μαζί κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει αυτό. Είπα τη λέξη δημοψήφισμα και ανατρίχιασα μια που έχουμε η Βρετανία, λέει ο πρόεδρο. Διευθυντή, Λάουρα Φερά. Ευχαριστώ πρόεδρε, καλημέρα κύριε επίτροπε. Σύντομα, πρόκειται να αρχίσουν οι κινήσεις για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για την διαφορά και το οργανωμένο εγκλήμα. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξή. Προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες όσον αφορά τους ελάχιστους κοινού κανόνες τόσο ώστε να εξασφαλίσει μια εναρμόνιση όσον αφορά τον ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος ή στο τι ορίζεται μαφιόζικου τύπου συμμορία. Και έτσι να μπορούμε να έχουμε λειτουργικότητα και επιχειρησιακή δυνατότητα του, Ευρωπαίου Σαγγελέα που θα πρέπει να εμπλακεί στην καταπολέμηση της απάτης της βάρος των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό ότι μόλις θα αρχίσει να λειτουργεί η υπηρεσία έχουμε το άρθρο 86 της συνθήκης που του απονέμει τη σχετική αρμοδιότητα για κάποια σοβαρά ε, διασυνοριακού χαρακτήρα εγκλήματα. Οπότε είπαμε ότι θα υπάρξει τότε η νομική βάση για να έχουμε κάποιους κοινού κανόνες κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, προτίθεστε να κατεβάσετε και προτάσει προτάσεις ούτως ώστε να έχουμε μια εναρμόνιση ε, για την περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και σε αυτό το τομέα έχουμε δράση οργανωμένων εγκληματιών εις βάρος των Ευρωπαίων. Τώρα όσον αφορά την διαφθορά, προτίθεστε να υπάρξουν κάποια όργανα, εργαλεία, μέσα παρακολούθησης και έτσι να μπορέσουμε να προλάβουμε ή να διώξουμε κάποιο είδου συστημικής φύσης ε, απάτη. Και σε επίπεδο πρόληψη. Επίσης να δούμε πώς θα συνεργαστεί με την Eurojust στο το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Γι' αυτό είναι πολύ θετικό το όσο συζητά τώρα το Συμβούλιο και προχωράει καλά το θέμα. Όσον αφορά την ε, ριζοσπαστικοποίηση στι φυλακές. Ε, πάρα πολύ σωστό ότι θα γίνει αυτή η διάσκεψη για την ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών. Και επίσης ελπίζω ότι θα υπάρξει θέληση να εστιάσουν προσοχή μας σε κάποια μέτρα σοφρονισμού εναλλακτικά της φυλάκησης. Πολύ συχνά και σε πολλές χώρες γίνεται κατάχρηση του σοφρονιστικού μέσου της κράτησης. Γι' αυτό και έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές. Όμως πολλέ φορέ οδηγούμεθα ακόμα και σε παραβίαση των δικαιωμάτων. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε κάπως τα δικαϊκά συστήματα και έτσι να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Τώρα για το Justice Scoreboard, τον πίνακα επιδόσεων στη δικαιοσύνη, ε, σε κάποια άλλη συζήτηση που ήσασταν κι εσείς, το είχαμε συζητήσει και είχαμε πει τι πιστεύετε όσον αφορά αυτό το πίνακα επιδόσεων, κυρίως για τα ποινικά. Και είχατε δείξει θετική στάση. Μετά συζήτησαμε τον κύριο Τίμερμα στη σχετική ακρόαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ο κύριος ε, Τίμερμαν ήταν λιγότερο θετικός. Δεν το βλέπετε τόσο εύκολο. Οπότε για πέστε μας, εσείς τι πρεσβεύετε τι θα κάνει η Επιτροπή. Είναι το να έχει ενιαία στάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θεμελιώδη δικαιώματα τώρα. Συμφωνώ με το όσα είπε η συνάδελφος Ινέτφελτ. Διότι χρειάζεται ένα σύστημα παρακολούθησης της κάθε χώρας όσον αφορά το τι κάνουν για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να επινοήσει ε, κάποια μέσα παρακολούθησης και αυτά να δρουν και σε επίπεδο πρόληψης. Ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε ένα κύκλο ερωτήσεων. Όπως είπαμε οι συντονιστές υπάρχει για τον καθόμενο διάλογο και συμφωνητών των πολιτικών ομάδων. Και αυτό έπρεπε να υποβάλουν ε, ερώτηση που οι πρώτοι συντονιστέ ε, εγώ φταίω. Έπρεπε να δώσω πρώτα πρώτα το λόγο. Και ο κύριο Νίτερ Μίλλερ και, οι άλλοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο τώρα. Ε, δεν είναι σωστό για αυτού, αδίκησα. Έπρεπε εκείνοι πρώτοι να ρωτήσουν. Οπότε, μήπω τώρα θέλουν να υποβάλουν τι ερωτήσει του, παρακαλώ σύντομα. Επαναλαμβάνω για τον διαρθρωμένο διάλογο. Άρα πήγε αυτό το θέμα να έχουμε μόνο τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Είναι ο κύριος Νίτερ Μίλλερ πρώτος και ο κύριος Μπόνι μετά. Νίτερ Μίλλερ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος κύριε Επίτροπε. Έχουμε συζητήσει πάρα, πολύ, πάρα πολλές φορές το θέμα της εκπαίδευσης ε, τον Ρωμά στην Ευρώπη. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιωθεί η κατάσταση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπονι, θέλετε να κάνετε την ερώτησή σας. Με συγχωρείτε, μία ερώτηση έχω μόνο. Γιατί καταλαβαίνουμε πως η προστασία των δεδομένων είναι βασικό θέμα και επίσης ε, χρειάζεται και μια οδηγία αλλά όταν ξεκινήσουμε την οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτική ζωή που αναφέρεται νομίζω στο ε, πακέτο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα πρέπει νομίζω να αρχίσουμε να την συζητάμε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, καλά τα πήγαμε. Νομίζω υπάρχει χρόνος να απαντήσετε, οπότε με την ησυχία σας. Έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε με την άνεσή σας. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα τσεχικά γιατί είναι η μητρική μου γλώσσα και έτσι θα μιλήσω πιο άνετα. Σας ευχαριστώ για όλα σας τα ερωτήματα. Πρώτον, κυρία Χολμάγερ, το ερώτημά σας για την Eurojust. Ρωτήσατε αν υπάρχει αναγκαιότητα να υποστηρίξουμε τη Eurojust και ως προς το προσωπικό της και ως προς τη χρηματοδότησή της γενικότερα Το έχω μελετήσει κι εγώ και έμαθα ότι αυτή τη στιγμή η νέα υπηρεσία ΕΠΟ σχεδιάζεται και σύμφωνα με τις συνθήκες φαίνεται ότι σήμερα η Eurojust δεν αρκεί. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και από την ΕΠΟ που θα αναλάβει επίσης κάποιο προσωπικό και κάποιες πληροφορίες από τη Eurojust. Όταν λοιπόν προετοιμάζεται η διοργάνωση της λειτουργίας της ΕΠΟ πρέπει να δούμε παράλληλα τι θα γίνει και με τη Eurojust. Δεν είναι λοιπόν αυτός ο μόνος λόγος για τον οποίο το θέμα θα συζητηθεί τους επόμενους μήνες. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη Eurojust και να την προωθήσουμε ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Και πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ χωρών μελών Ευρωπόλ και Eurojust. Ταυτόχρονα η Eurojust πρέπει να συνεννοηθεί με τρίτες χώρες που, από όπου προέρχονται πολλοί εγκληματίες. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση και σε τρίτες χώρες. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους τα καθήκοντα της Eurojust πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο. Είμαι πεπισμένη ότι η Eurojust δεν μπορεί να λειτουργήσει ως έχει. Πρέπει να την προωθήσουμε γιατί υπάρχει και το νέο πρόγραμμα για την ασφάλεια και πρέπει να εναρμονίσουμε ή να υπάρξει συνεργασία, να συνδυάσουμε τη δουλειά της Eurojust με την καινούργια υπηρεσία ΕΠΟ. Τώρα λοιπόν. Γι' αυτό το ΕΠΟ δηλαδή την υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Έχει συμφωνηθεί, ήταν πολύ σημαντική δουλειά της προηγούμενης Κομισιόν θα οριστούν ειδικοί εισαγγελείς και σε κάθε περίπτωση σε κάθε λέω περίπτωση λέω όποτε χρειάζεται συνεργασία που δε, όπου δεν φτάνει δηλαδή το απλό εθνικό επίπεδο θα γίνει θα υπάρξει μια ειδική δικαστική διαδικασία η υπηρεσία αυτή η ε, ΕΠΟ λοιπόν θα ελέγχεται και αυτή, θα εποπτεύεται, αλλά είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε την ποιότητα των δικαστικών συστημάτων στις χώρες μέλη. Υπάρχουν μερικοί δείκτες, αλλά δεν ξέρω αν δεν, μήπως δεν είναι παραπλανητικοί μερικοί από αυτούς. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε να συγκρίνουμε τα στατιστικά στοιχεία της Όλαφ όπου υπάρχουν περιπτώσεις διαπιστωμένης απάτης και μπορούμε επίσης να δούμε πόσες από τις διαπιστωμένες απάτες έχουν εκδικαστεί στα κράτη-μέλη. Μπορούμε δηλαδή να συγκρίνουμε τα στατιστικά στοιχεία περιπτώσεων που έχουν καταλήξει επιτυχώς, διεκπαιρεωθεί επιτυχώς. Είναι και αυτός ένας λόγος για την ύπαρξη της ΕΠΟ, με τα ίδια όμως κριτήρια σε όλες τις χώρες μέλη. Δεν θέλω να κατηγορήσω καμία συγκεκριμένα, αλλά ξέρω ότι μερικές φορές υπάρχουν καταχρήσεις κατάφορες γιατί σε μερικές χώρες δεν είναι εύκολη η εκδίκαση ή η απλή διερεύνηση περιπτώσεων απάτης. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε μεγαλύτερη φρόνηση σε χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη εισρωή ενωσιακών κεφαλαίων. Υπάρχουν ερωτήσεις και για τον ασφαλή λιμένα, <clears throat> όπως είπε η κυρία Χόλμαγερ, για το σύστημα επιτήρησης του, αν κατάλαβα καλά λέει η Επίτροπος. Έχουμε δημοσιεύσει 13 συστάσεις 11 από αυτές αφορούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδαμένων. Οι συστάσεις αυτές αφορούν και τρίτες χώρες. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε και για αυτές. Τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση της συμφωνίας με το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε θέσει συγκεκριμένους και σαφείς όρους ως προς το πώς εξοφίκιο θα γίνεται ο έλεγχος των όρων λειτουργίας. Και υπάρχουν και ειδικέ ρήτρες για τους ελέγχους για συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και επίσης θα υπάρξει ειδική ενισχυμένη συνεργασία με τις αρχές που ασχολούνται με την, που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων παραβίασης. Είμαι σίγουρη ότι οι 11 αυτές τάσεις από τις 13 θα τις δεχτείτε κι εσείς και τις δεχτήκατε μάλλον ήδη και γι' αυτό νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο όπως σας είπα αυτές οι 13 συστάσεις έχουν υποβληθεί και οι δύο εναπομένουσες αφορούν τη χρήση προσωπικών δεδομένων από υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτές οι δύο τελευταίες συστάσεις βέβαια είναι πολιτικά πολύ ευαίσθητες. Όποιος ενδιαφέρεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να ενδιαφερθεί και για αυτές τις δύο συστάσεις που είναι τόσο σημαντικές. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε τελικά να τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τους συγκεκριμένους όρους μέχρι το τέλος Μαΐου. Δεν θα μπορέσουμε. Αναμένω λοιπόν στη Ρήγα, στην υπουργική διάσκεψη, μια ειδική διάσκεψη μεταξύ ΙΠΑ και, Ενωμένων και Ένωσης, ότι εκεί θα, μπορέσω να, θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την κατάληξη αυτών των διαπραγματεύσεων και μετά αργότερα μαζί με τον κύριο Τίμερμανς και άλλους επιτρόπους ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε κατά πόσον όλα αυτά που συμφωνήθηκαν αρκούν. Άλλο θέμα είναι κατά πόσον το safe harbor πρέπει να ακυρωθεί ή όχι. Ναι, συζητιέται και αυτό, συζητιέται. Οι εγγυήσεις της αμερικανικής πλευράς εάν αποδειχθούν ανεπαρκείς τότε το θέμα θα ξανατεθεί και τότε θα δούμε αν συνεχίσουμε να συζητούμε την αρχή του Safe Harbor ή εάν πρέπει να ακυρωθεί. Για να τα πω λίγο απλά, ίσως δεν πρέπει να έχουμε πολύ ψηλέ προσδοκίες. Μπορεί κάτι να συμφέρει το εμπόριο και όσοι το εκπροσωπούν φοβούνται για την ακύρωση του Safe Harbor. Δεν πρέπει όμως να καταλήξουμε σε παγίδες. Αν κάποιο σύστημα δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, τότε θα ταχθώ κατά του. Πρέπει να περιμένουμε όμως λίγο παραπάνω χρόνο και μέχρι τα τέλη του Ιουνίου ελπίζω οι διαπραγματεύσεις αυτές να έχουν καταλήξει και τότε θα συζητηθεί το θέμα με τους επιτρό... μεταξύ επιτρόπων και θα σας ενημερώσω. Δεν μίλησε κανείς για τη γενικότερη συμφωνία όμως ίσως τα πράγματα να είναι πιο θετικά από ό,τι φαίνεται. Έχουμε ένα πρώτο κείμενο, ένα πρόχειρο κείμενο, ένα προσχέδιο και μόνο ένα ακόμη πρόβλημα έχει παραμείνει. Τα δεδομένα που θα μεταφερθούν από το ομοσπονδιακό σε πολιτιακό επίπεδο. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτή. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει το ομοσπονδιακό επίπεδο να είναι υπεύθυνο και να είναι σαφής η όροι με τους οποίους θα γίνει αυτή η μεταφορά. Προσπαθούμε να πετύχουμε σαφή συμφωνία σε περίπτωση εφόσον υπάρχουν μόνο μερικές υποθέσεις όπου θα χρειαστεί αυτή η μεταφορά αλλά και σε αυτές τις ίδιες περιπτώσεις θα χρειαστεί. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών θα συζητήσει το θέμα και τότε θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για να ζητήσουν οι Ευρωπαίοι νομική προστασία. Ξέρετε ότι για Ευρωπαίους είναι τελείως απαραίτητο να χορηγηθεί τέτοια νομική προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπάθησα να απαντήσω όσο μπορούσα για το Safe Harbor, τώρα τα θεμελιώδη δικαιώματα και η Ρωμά ας πούμε. Έχουμε λάβει εθνικά προγράμματα για αυτό το θέμα και υπάρχουν μερικά στοιχεία πρωτότυπα καινοτομίες ας πούμε η αναγκαιότητα να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για να προωθηθεί η ολοκλήρωση και συνεργασία των Ρωμά με την κοινωνία στην οποία ζουν. Αυτά είναι πράγματα που συμπεριλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα που γενικά τονίζουν τη σημασία των τοπικών αρχών και τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρές καινοτομίες και πρωτοτυπίες που προτείνονται όπως η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης για κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες όπως στη Ρουμανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί ανέχειας γενικότερα αλλά μεταξύ των πτωχοτέρων μια πλειοψηφία Ρωμά. Ξέρουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης τους στη Ρωμανία τους αναγκάζουν να φύγουν από τη χώρα σε άλλες ευρωπαϊκές και μετά τίθενται προβλήματα ιδιαίτερα στη Γαλλία και τη Σουηδία από τους Ρωμά και η Ρουμανία προσπαθεί να διαπραγματευτεί κάποιο είδους συνεργασία. Δεν είναι ενωσιακό θέμα βέβαια, αλλά πρέπει να σας το πω διότι ε, πρόκειται για διμερεί θέματα μεταξύ χωρών μελών και αφορούν τους Ρωμά, γι' αυτό τα αναφέρω. Οι στρατηγικές, αυτά τα προγράμματα αν εφαρμοστούν μπορεί να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Από τα μέτρα που συζητάει η Κομισιόν μπορεί να ξέρετε ότι δημοσιεύσαμε μία σύσταση σε πέντε χώρες μέλη συγκεκριμένα για τους Ρωμά και την ε, εκπαίδευσή τους στα δημοτικά και οι συστάσεις αυτές αφορούν την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα εάν δεν απατώμε, όχι, όχι την Ελλάδα, τη Βουλγαρία. Αυτές είναι οι χώρες λοιπόν που έχουν λάβει συστάσεις. Τις υποβάλαμε πρόσφατα. Μετά υπήρχε ένα άλλο θέμα για τους Ρωμά στα σχολεία έχω τη δυνατότητα να απαιτήσω την εφαρμογή την ε, παρεμπόδιση της τοποθέτησης Ρωμά, παιδιών Ρωμά σε σχολεία για διανοητικός αναπήρους γιατί καμία μελέτη δεν έχει ποτέ αποδείξει ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο και το ίδιο ενδιαφέρουσα είναι ενδιαφέρον είναι το θέμα των ρατσιστικών επιθέσεων. Πάλι καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει ότι όντως ένα τρίτο των Ρωμά είναι διανοητικός ανάπηροι. Αυτά είναι ανοησίες. Υπάρχει λοιπόν η αναγκαιότητα νέου, νέας διάγνωσης για να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και να διορθωθούν τα ποσοστά. 35% στην Τσεχία των παιδιών Ρωμά φοιτούν σε σχολεία για διανοητικώς καθυστερημένους. Και ήταν η πρώτη χώρα για την οποία στείλαμε επιστολή από την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Συνέχισε η ανταλλαγή επιστολών και σε λίγο θα κάνουμε μία δε δικαιολογημένη γνωμοδότηση. του χρόνου πια βέβαια από την 1η Ιανουαρίου. Τα αποτελέσματα, πρώτα αποτελέσματα λοιπόν θα φανούν το Σεπτέμβριο του 2016. Προτιμώ λοιπόν να ζητήσω δέσμευση από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας ότι φέτος η διάγνωση για τα ποσοστά παιδιών με πνευματικές αναπηρίες θα αλλάξει. Η πραγματική αριθμή θα φανούν φέτος τον Σεπτέμβριο. Αριθμοί που θα δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Αυτό είναι καλύτερη μέθοδος νομίζω για μένα από ότι να κάνουμε μία απλώς επίσημη δε δικαιολογημένη γνωμοδότηση. Αυτό βέβαια θα ελκύσει και την προσοχή, θα ελκούσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά δεν είναι η προσέγγιση που προτιμώ γιατί και σε άλλες χώρες υπάρχουν προβλήματα με την παιδεία των Ρωμά. Mm. Για τους ΛΟΑΕΔ ήταν δύο τα ερωτήματα, θα τα απαντήσω μαζί. Προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει πρόβλημα εδώ. Αλλά το συζητώ με τους άλλους επιτρόπους. Γιατί είναι πρόβλημα να προετοιμαστεί το πρόγραμμα φέτος. Υπάρχουν τρεις προτεραιότητες. Η μία είναι να καταλήξει η νομοθεσία που αφορά τους ΛΟΑΕΔ και εννοώ την ίση μεταχείριση, την οδηγία. Δεύτερον, πρέπει να παρακολουθήσουμε τι προβλήματα υπάρχουν στα κράτη-μέλη προς αυτό και πρέπει να αναλύσουμε, να αναλύσουμε τα στοιχεία για να δούμε πού θα ήταν πιο αποτελεσματικό να υπάρξει νομοθεσία και που ήταν καλύτερο απλώς να υπάρξει κάποια πληροφόρηση, καμπάνια πληροφόρησης μέσω μη κυβερνητικών ίσως οργανώσεων. Αυτό τον καιρό εξετάζω την αναθεώρηση της χρήσης 52 εκατομμυρίων από τη Γενική Διεύθυνση Δικαστικών και νομίζω ότι η κοινωνία των πολιτών θα εγκρίνει τα μέτρα αυτά γιατί η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να κάνουν πολλά αν έχουν σωστά στοχευμένες καμπάνιες. Για το πρόγραμμα δράσης για τους ΛΟΑΕΔ λοιπόν αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. να καταστρώσουμε την πολιτική μας από φέτος θεωρητικά τουλάχιστον και να γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ημών και ημών με τη Σοφή, με την κυρία Λούνετσεκ μπορούμε να δούμε αν αυτό θα προχωρήσει τα πράγματα ή όχι. Αργότερα θα διαπραγματευθώ μεταξύ επιτρόπων το θέμα Πρέπει βέβαια να αποσαφηνίσουμε αν πρόκειται πράγματι για οδικό χάρτη ή πρόγραμμα δράσης. Δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι για την ορολογία, αλλά συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Η υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βιέννη σε λίγο θα αλλάξει ηγεσία και προσβλέπω και σε αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για το Ιρλανδικό δημοψήφισμα. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό. Μετά για την περίπτωση Σρέμπου. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έλεγε η ερώτηση, αλλά βιαζόμαστε αυτή τη στιγμή, θέλουμε να ενδυναμώσουμε το safe harbor και να καθορίσουμε εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων για να μην επηρεάσουμε βέβαια τη δικαστική διαδικασία αλλά για να δείξουμε ότι η Κομισιόν δουλεύει και μάλιστα πολύ σκληρά και μπορούμε να αναμένουμε βελτίωση της κατάστασης. Περιμένουμε τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα στις 24 Ιουνίου. Μέχρι τότε τότε θα δούμε εάν θα συνεχίσει ή όχι το safe harbor και θα συνεχίσει μόνον με πολύ ενδυναμωμένο τρόπο μόνο όσο για την προστασία των δεδομένων και τον κανονισμό υπήρχε το θέμα το ερώτημα του κατά πόσον είναι ακόμη δέσμοι μαζί με την οδηγία για την αστυνομία ναι μικρή θα είναι η αλλαγή και η μετατόπιση για τον κανονισμό αναμένουμε αναμένουμε λέγω την Γενική Προσέγγιση του Συμβουλίου τον Ιούνιο και οι διαπραγματεύσεις θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό νομίζω γιατί είναι πολλά τα θέματα και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα περιφερειακά και περιθωριακά προβλήματα για να ασχοληθούμε με τα βασικά. Ελπίζω μετά τις 24 Ιουνίου να γίνει ο πρώτος τριμερής διάλογος όπου θα παρίσταμε και εγώ μαζί με τους υπουργούς και αναμένω και εκπροσώπηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά και ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα συνεχίσει στις 16, από τις 16 Ιουλίου και μετά. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα μόλις εγκρίνει το πράγμα το Συμβούλιο. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μας διότι μας βοηθάτε πολύ στις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Όσο για την οδηγία για την αστυνομία. Τον Ιούνιο αναμένουμε μια μερική προσέγγιση και το δεύτερο εξάμεινο επί Λουξεμβουργικής Προεδρίας αναμένουμε την τελική έγκριση στο Συμβούλιο. Ίσως γνωρίζετε ότι τον Ιανουάριο είχαμε το δευτερεύον θέμα, ένα δευτερεύον θέμα που αφορούσε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και γνωρίζει ο εισηγητής πως προσπαθήσαμε να το διατηρήσουμε ανέπαφο και όσον αφορά την οδηγία και όσον αφορά τον κανονισμό και ταυτόχρονα εξηγήσαμε την θέση μας ε, στη Γερμανία και στις άλλες χώρες που έθεσαν το ζήτημα και νομίζω πως ε, καταλήξαμε σε κάποιες ε, ικανοποιητικές λύσεις χρησιμοποιώντας κάποια ευελιξία για να διατηρήσουμε το πεδίο εφαρμογής. Τώρα έχω γράψει κάτι εδώ πέρα και δεν βγάζω τα γραμματά μου. Λοιπόν, αφορά την ερώτηση της Σόφι ε, Νιτφέλτ. Κάποια πράγματα τα έχω απαντήσει, αλλά τώρα δεν μπορώ να απαντήσω για την αξιολόγηση της καταπολέμησης ε, της τρομοκρατίας και το αν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Βεβαίως, ε, η ατζέντα της ασφαλείας θα αξιολογείται συνεχώς και θα είναι αντικείμενο δικό μας του Κοινοβουλίου και της ε, κοινή γνώμης οπωσδήποτε. Για την οδηγία κατά των διακρίσεων φοβούμε λίγο. Θέλω να λέω θελικά πράγματα, αλλά εδώ πέρα η κατάσταση είναι κάπως πιο περίπλοκη. Υπάρχουν δύο προβλήματα λοιπόν με αυτή την οδηγία. Κανένα κράτος μέλος δεν λέει πως η οδηγία είναι κακή, διότι δεν χρειάζεται. Η οδηγία αυτή αφορά ένα βασικό πράγμα, τη μη διακριτική μεταχείριση στον τομέα των υπηρεσιών για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά ε, το θέμα είναι η επίδραση στον προπολογισμό. Με απλά λόγια πρόσβαση για ανάπηρους στα κτίρια για άτομα με ε, καρεκλάκια αναπηρικά και βεβαίως όταν μιλάμε για οδηγία είναι κάτι το οριζόντιο και δεν ε, είναι πραγματικά ένας συγκεκριμένος αρμόδιος σε κάποια κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Αλλά παρόλα αυτά σας υπόσχομαι πως θα πιέσουμε για να περάσει αυτή η οδηγία. Δεν θα αναφέρω τώρα ποια κράτη-μέλη μου είπαν ότι έχουν πρόβλημα με αυτή την οδηγία. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί μέχρι το δεύτερο εξάμεινο του έτους για να έχουμε καλύτερη στήριξη από τα κράτη-μέλη. Τώρα για την Ουγγαρία πρέπει να πω πως ε, παρακολουθούμε την κατάσταση στενά. Το τελευταίο θέμα αυτό της θανατικής ποινής πραγματικά δηλαδή ήταν τελευταία στα αγώνα. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Μετά λάβαμε τις εξηγήσεις ότι δεν το λέγαν σοβαρά Απλά ε, είπαν κάτι για να το πούνε. Ε, μα αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να δούμε την συστηματική παραβίαση των συνθήκων στην Ουγγαρία. Συνεχώς ε, πάντα εμφανίζεται κάτι ε, που είναι παραβίαση των συνθήκων και μετά υπάρχει μια λύση που είναι να πηγαίνουμε στα δικαστήρια και μετά η Ουγγαρία λαμβάνει κάποια μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση. Μετά είχαμε ΜΚΟ που έπαιρναν λεφτά από ε, Νορβηγούς και πήγα εκεί πέρα να δω την ε, κατάσταση και το πώς ε, έχει το κλίμα το δημοκρατικό στην χώρα αυτή όσο μπορεί να κρίνει κανείς με μια επίσκεψη και μου είπαν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ όπως υπήρχαν αστυνομικές ε, έφοδοι και φοβόταν το τι θα γίνει και μετά αφού έφυγα ε, το θέμα λύθηκε γιατί το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ των ΜΚΟ. Οπότε στην Ουγγαρία κάτι συμβαίνει και μετά λύνεται. Και πάντα έτσι πάει το πράγμα. Και εγώ και ο Φράντ Τίμερμαντ έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα αυτό, για την κατάσταση της δημοκρατίας σε όλες ε, τις ε, χώρες ε, τις οποίες πρέπει να μεταχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε παρακολουθούμε την κατάσταση και μόλις γίνει αφόρητη θα δράσουμε και θα δημιουργηθεί, θα ξεκινήσει ο μηχανισμός όπως αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν μπορώ να σας πω πότε θα γίνει κάτι τέτοιο γιατί εξαρτάται από το τι γίνεται στην Ουγγαρία και στις άλλες ε, χώρες. Και εδώ πέρα πρέπει να πω πως ε, μια διαδικασία επί παραβάση είναι κάτι το αναγκαίο για την Κομισιόν και στέλνει και ένα μήνυμα σε άλλες χώρες. Οπότε είναι ζήτημα ακριβώς της κατάλληλης ε, πολιτικής στιγμής. η προσχώρηση στην ε, ε, ΕΣΔΑ και εμένα έναν σε έκπληξη η απόφαση του δικαστηρίου μας καθυστέρησε και σε άλλα πράγματα όπως η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών. Περιμένουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου. Δύο λύσεις υπάρχουν λοιπόν. Δεν κάνω εγώ την ανάλυση αυτή, δεν είναι η δικιά μου γενική διεύθυνση, αλλά αναμένουμε τα αποτελέσματα και δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Είτε θα το δεχτούμε και δεν θα γίνουν άλλες απόπειρες ή θα ξαναγράψουμε το σχέδιο σύμβασης προσχώρησης και θα ξαναξεκινήσει η πολύπλοκη διαδικασία της κύρωσης. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν αν είναι απαραίτητο ή όχι. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Και σας λέω ότι θα ε, καταβάλω κάθε προσπάθεια. Τώρα, όσον αφορά την ε, έκθεση για την διαφθορά. είναι περισσότερο ένα ερώτημα προς την ε, κυρία Γιούρκεβα. Εγώ κυρίως ε, το βλέπω μέσω της Ευρωπαϊκής ε, εισαγγελία. Εάν εναρμονίσουμε τα ποινικά δικαιώματα, η Ευρώπη έχει νομίζω κάποιες αρμοδιότητες τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε. Οπότε θα προσπαθήσουμε να αναρμονίσουμε τους όρους τρομοκρατία και ξένος μαχητής ε, στον τομέα της ασφάλειας. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ε, το κοιτάει το ζήτημα σε συνεργασία μαζί μας. Ξέρετε πως και ο ΙΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, έχουν έναν ορισμό της τρομοκρατίας που περιλαμβάνει και το φαινόμενο των ξένων μαχητών. Επίσης γνωρίζετε πως σε κάποια κράτη-μέλη ο ορισμός στον ποινικό κώδικα δεν αρκεί. Εάν ένας νεαρός ε, που ζει δίπλα σας λέει πως τα μαζεύει για τη Συρία, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία να τον σταματήσετε. Δεν είναι ποινικό αδίκημα να προετοιμάζει κανείς ε, να προετοιμάζεται για τρομοκρατικές πράξεις. Σημαντικό αυτό λοιπόν η εναρμόνιση και στο πλαίσιο της έγκαινης και της ελεύθερης ε, μετακίνησης. Όσον αφορά λοιπόν την εναρμόνιση αυτή των ποινικών δικημάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ελπίζω ότι η ερμηνεία το, της ε, ζημιάς των οικονομικών συμφερόντων της ε, κοινότητας ε, θα ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί η ερμηνεία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Την παρακολούθηση της Ουγγαρίας, τα ΙΠΑ, Ρωμά, εκπαίδευση, η ηλεκτρονική ιδιωτική ζωή θα συνεχίσουμε. Δεν έχω τίποτα πιο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς αγαπητοί συνάδελφοι ότι γι' αυτόν τουλάχιστον το διαθρωμένο διάλογο είχαμε αρκετό χρόνο και απαντήθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Και πιστεύω πως και εσείς κυρία Πίτροπε, θα συμφωνήσετε πως ε, δεν βιαστήκατε να μας δώσετε απαντήσεις και είχατε όλο το χρόνο που χρειαζόταν. Αυτό λοιπόν είναι μια επιτυχία. Αυτό όμως που μας ελειπεί είναι ότι οι άλλοι συνάδελφοί σας δεν κατάφεραν να έρθουν. Και αυτό είναι κάτι που θα συζητήσω με τους συντονιστές, θα το πότε δηλαδή θα δούμε τους επιτρόπους Τίμερμανς και Αβραμόπουλο στα πλαίσια του διαθρωμένου διαλόγου. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι το πρόγραμμα εργασίας για το 2016 και σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές. Θα μπορούσατε και εσείς να μου προτείνετε κάποιες δικές σας ιδέες. Έχω τις ε, προτάσεις του επιτελείου μου. Νομίζω όμως πως ε, πρέπει να το αναλύσουμε. διότι με ανησυχεί αυτό και έχω ακούσει πως ε, δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητές οι εναλλακτικέ μέθοδοι σοφρονισμού. Οι πολίτες θέλουν να βλέπουν τους ε, κακοποιούς στις φυλακές και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήμουν ευγνώμων για όλες τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω ότι μετά το τέλος του διαρθρωμένου διαλόγου θα ε, στείλουμε και γραπτά τις προτάσεις αφού αυτές εγκριθούν από τη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών. Να σας πω τώρα πως ε, συνοψίζοντας η Επίτροπος ε, κατέστησε σε αμφές πως θα συμμετέχουν όλα τα μέλη. Και εγώ σημείωσα τα κύρια σημεία που συζητήσαμε. Καταρχάς η Eurojust και το θέμα του προσωπικού, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η συμβατότητα του Safe Harbor με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στρατηγική για τους Ρωμά και τους ΛΟΑΔ, ομαλή λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταρρύθμιση, οριζόντια οδηγία και να προσθέσω και εγώ επίτροπε ότι η συζήτηση για το Safe Harbor άρχισε το 2013 σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και είναι κάτι που συνεχίζουμε να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουμε δηλαδή περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι ήρθατε στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια και μας ενημερώσατε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ξανά για τις απαντήσεις σας. Μας βοηθήσατε πολύ και εγώ θα ήθελα να ε, σας ευχαριστήσω. Συνάδελφοι, να πω, ιδιαίτερα για όσους ήρθαν πριν από λίγο, πως έχουμε κάποιες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη. Πριν αναλύσουμε την κατάσταση στη Μεσόγειο, θα συζητήσουμε το σημείο 8 το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το 2015 και την απάντηση στις ε, μετανασκευτικές πιέσεις. Θα έχουμε μία παρουσίαση από τον Ματία Ρούτε, Γενικό Διευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος μόλις έφτασε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 23 Απριλίου το Συμβούλιο εξέδωσε μία δήλωση για κάποια μέτρα που θα ληφθούν ως απάντηση της κρίσης, στην κρίση στη Μεσόγειο. Κάποια από τα μέτρα αυτά ερμηνεύτηκαν ε, δημοσιονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2015. Και συγκεκριμένες προτάσεις για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα μας παρουσιάζει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού του 2015 και θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Ρούτε για να μας ενημερώσει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ήρθα σήμερα για να σας ενημερώσω σχετικά με τις ε, ουσιώδεις λεπτομέρειες του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2015. Όπως θα γνωρίζετε, ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος θα ενημερώσει αύριο το Κοινοβούλιο ότι εμείς θα εφαρμόσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση και θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αύριο όμως, δυστυχώς, δεν μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό σήμερα. Σήμερα θα σας μιλήσω για πόρους. Και στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γεγονότα στην Μεσόγειο, τα πρόσφατα γεγονότα στη Μεσόγειο. 90 εκατομμύρια ε, πιστώσεις και περίπου 60-70 ε, εκατομμύρια σε πληρωμές είναι τα κονδύλια. Καταρχάς σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό της Frontex κατά 27 εκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις κοινέ επιχειρήσεις Τρίτων και Ποσειδώνας, για τους επόμενους μήνες του 2015. Επίσης, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την εναέρια και θαλάσσια επιτήρηση σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος για να το συνδυάσουμε και με το πρόγραμμα Mare Nostrum. Το 2016 οι ανάγκες θα καλυφθούν από τον προπολογισμό για το αντίστοιχο έτος. Έπειτα, έχουμε προτείνει αύξηση πόρων για το Ταμείο Μετανάστευσης και Ένταξης. 57 εκατομμύρια δεσμεύσεις και 45,6 εκατομμύρια πληρωμές και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας επίσης με ...4,5 και 5 εκατομμύρια αντίστοιχα. από τα χρήματα αυτά, τα 25 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για συστήματα έκτακτης ε, ανάγκης στα προγράμματα της πρώτης γραμμής, αν και δεν μου αρέσει αυτή η διατύπωση. Για περιοχές λοιπόν οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αυξημένο μεταναστευτικό κύμα στα πλαίσια της ε, επιχείρησης Ποσειδών. Αυτό που θα κάνουμε δηλαδή είναι να ενισχύσουμε καταρχάς τις δυνατότητες υποδοχής ε, κατά την άφηξη, ε, για την στέγαση, για την ιατρική εξέταση και την μεταφορά των μεταναστών και τη σύντηση επίσης. Τα υπόλοιπα 25 εκατομμύρια θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο μεταγκατάστασης. Αυτό που έχει προτείνει ο Επίτροπος δηλαδή πριν από μόλις δύο εβδομάδες για περίπου 2.000 νέες θέσεις μεταγκατάστασης σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως θα δείτε, αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει για τις ε, λεπτομέρειες αυτών των ε, θέσεων μετεγκατάστασης. Επίσης, 7 επιπλέον εκατομμύρια στα πλαίσια του ΆΜΕΦ θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν το πρόγραμμα περιφερειακής προστασίας και αυτό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για τη μετανάστευση, για τις χώρες προέλευσης, χώρες διαμετακόμισης, χώρες προορισμού. και θα μας βοηθήσει να καλύψουμε τις πρόσθετες ανάγκες που θα προκύψουν σε τρίτες χώρες. Και τρίτον, έχουμε προτείνει αύξηση του προσωπικού των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Φυσικά η Frontex έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Γι' αυτό έχουμε προτείνει δημιουργία 16 επιπλέον νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, Αυτές οι θέσεις θα ασχοληθούν με την ε, ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, τρεις επιπλέον θέσεις για την Ευρωπόλ και τέσσερις επιπλέον θέσεις προσωπικού για την ε, ΕΑΣΟ. 16 λοιπόν, 3 και 4. Επίσης, έχουμε εντοπίσει μη χρησιμοποιημένες επιστώσεις προϋπολογισμού σε άλλους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα ποσά ανέρχονται στα 75,8 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων, άρα δεν χρειαζόμαστε επιπλέον πιστώσεις πληρωμών. Αυτά προς το παρόν. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας με τα χαράς. Σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Δεν ξέρω πόσες φορές σας είπα για τις συναντήσεις των συντονιστών. Έχει λάβει επικές διαστάσει. Το αποφασίσαμε όλα εκεί πέρα γιατί μεταξύ άλλων τώρα αυτό που θέλω να, να δούμε είναι τι θα γίνει όσον αφορά ε, κάποια γνωμοδότηση για τον διορθωτικό προπολογισμό, να ορίσουμε κάποιον ε, εισηγητή. Να δούμε σήμερα. Περιθούν όλα και να δούμε προς το παρόν από εσά τι μπορούμε να μάθουμε. Σύμφωνα με όσο μας είπε η κυρία Ρούτα. Ο κ. πρέπει είναι ο πιο έμπειρος συνάδελφος υπό αυτόν. Ζεράρ, εσύ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι βέβαιο. ότι μακρά θητεία σημαίνει υψηλή ποιότητα. Αλλά τόσο πάνω σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να σας πω ότι θεωρώ, θεωρώ ότι θα υπάρξει προπολογισμός. Γιατί όντως χρειαζόμαστε επιπλέον πόρους. Αυτό απλώ να είναι η αρχή της διαδρομής. Αλλά έχω κάποιες ερωτησούλες, ε, κύριε γενική Πρώτον, για τη Frontex. Βλέπω ότι προτείνεται αύξηση κατά εκατομμύρια. Και λέτε και ότι έτσι θα τριπλασιαστεί η δύναμη της Frontex για το Τρίτον και για το Ποσειδόν. Σύμφωνα με φρέσκες πληροφορίες μαθαίνουμε ότι μέχρι τώρα έχουν εκταμιευθεί 3 εκατομμύρια μηνιαίως για αυτές τις επιχειρήσεις. Εσείς μιλάτε τώρα για 7. Αλλά 3 επί 3 κάνει 9. 6 επί 7 πάει 42, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω που, που, που είναι όλα αυτά τα οποία σας λέω, αλλά πού είναι όλα αυτά τα οποία λέτε. Α, λέτε για τριπλασιασμό της προοικοδότησης της ε, Frontex για τις επιχείρησεις τρίτων και υποσύδων. Πού κάνω λάθος. Για πέστε μου. Επίσης, είναι πάρα πολύ ε, θετικό το ότι ε, θα πάτε σε τα 57 εκατομμύρια αύξηση της προϋποδότησης του ΑΜΕΦ και μεταξύ αυτών θα έχουμε 7 εκατομμύρια τα οποία θα αφορούν την ενίσχυση των προγραμμάτων για Βόρεια Αφρική και Κέρατος Αφρικής. Αλλά από την άλλη μεριά, τα 7 εκατομμύρια είναι φραγκοδίφραγκα γιατί είναι τεράστιες οι προκλήσεις. Πού θα πάνε τα 7 εκατομμύρια, σε ποιον, για να κάνει τι. Για κοιτάξτε να δείτε πόσο ε, απίστευτε είναι οι ροέ οι μεταναστευτικέ. Γι' αυτό και σε την αστεία αυτά τα ποσά και θα πρέπει να το δούμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν ξέρω καν τι διαστάσει του. Τρίτον, για τι θέσει, την αύξηση των θέσεων των ε, υπαλλήλων. Καλά αυτά είναι και τις εκτόπιση των προπολογισμών. Πώ αυτό συνάδει με τον γενικό κανόνα της μείωσης του 5% στα πλαίσια των πολιτών ε, προοπτικών και λοιπά για θεσμικό όργανα και υπηρεσίες γιατί αφού θα αυξήσετε στις δικές σας υπηρεσίες τους υπαλλήλους τότε θα πρέπει να κόψετε ένα σωρό αλλού άρα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό άλλο όσον αφορά την κατανομή αυτών των θέσεων είπατε 16 θέσεις για τη Frontex να κάνουν τι προβλέπετε βλέπω εδώ στο έγγραφο ενίσχυση του ρόλου της Frontex όσον αφορά την οργάνωση των επιστροφών, επαναπατρισμών κλπ. Άρα τι να κάνουν οι 16 ακριβώς στη Frontex. Επίσης, οι άλλες τέσσερις θέσεις, τι καλά δεν είναι και τόσο τρομερή αύξηση όσον αφορά ε, το, την καταγραφή στο Μητρό, τη λήψη αποτυπωμάτων κλπ. Δεν έχω δει τον Και λέτε εδώ στα γαλλικά για την διακοπή των, των ροών και των διαδρομών αυτών των λαθρομεταναστών. Αυτό όμω δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο τη υπηρεσία ταχείας ταχεία αντίδραση. Δεν είναι πολύ σαφή όλα αυτά, αν μου επιτρέπετε. Γι' αυτό και θα σας ρωτήσω προς διευκρίνηση. Πρόεδρος. Όπως έλεγα κύριε Ντεπρέ, έχετε μεγάλη εμπειρία στον προϋπολογισμό και μας βοηθάει αυτό πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον κύριο Ντεπρέ. Ε, κύριε Ρούτε, ίσως για να μας βοηθήσετε να το κατανοήσουμε καλύτερα. Θα μπορούσατε να μας πείτε αυτή τη στιγμή ποια είναι τα μηνύα έξοδα, καταρχάς για τη Frontex, έπειτα για το, τα προγράμματα τρίτων και ποσειδών και τρίτων για την ΕΑΣΟ και η αλλαγή του προϋπολογισμού, τι θα σημαίνει μελλοντικά για αυτά τα τρία προγράμματα. και για την ε, Frontex και για την ΆΣΟ και για τα προγράμματα Τρίτων και Ποσειδών επίσης. Θα ήθελα να μάθω τι προσωπικό έχουν αυτή τη στιγμή. Και Τρίτων και Ποσειδών, αυτά τα δύο προγράμματα, εάν αυξηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού, είτε τριπλασιαστούν είτε όχι, τι θα γίνει, πού θα πάνε αυτά τα κονδύλια. Και ε, ε έχω την εντύπωση ότι μέχρι τώρα χρειάστηκε περισσότερο προσωπικό και περισσότερα κονδύλια, γιατί δυσκολεύονται πάρα πολύ τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το πακέτο για το άσυλο. Όμως από φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε ένα νέο πακέτο για το άσυλο και αυτό θα σημαίνει ακόμα περισσότερη δουλειά για τα κράτη-μέλη. Και Χρειάζεται λοιπόν να εφαρμοστεί το πακέτο αυτό όσο το δυνατόν ομαλότερα από όλα τα κράτη-μέλη και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επιπλέον, σχετικά με την επανεγκατάσταση, θα ήθελα να ρωτήσω πού βρισκόμαστε δεδομένων των μέσων που έχουμε αυτή τη στιγμή και σε πόρους και σε προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ, Μπίργκη. Την κυρία Χολμάιρ έχει το λόγο. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, εφαρμογή του πακέτου για το άσυλο. οι απόψεις από τα κράτη-μέλη διαφέρουν αρκετά. Την 1η Ιουλίου θα εφαρμοστεί το νέο πακέτο για το άσυλο και η εντύπωση που αποκομίζω από ορισμένα κράτη-μέλη είναι ότι δυσκολεύονται ως προς την εφαρμογή. Και επίσης άλλα κράτη-μέλη έχουν αρκετά διαφορετικές απόψεις σχετικά με το όλο πακέτο. Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω εσάς, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέση να έχει μια γενική εικόνα του τι γίνεται στα κράτη-μέλη, όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη για την ε, εφαρμογή ενώ των ελάχιστων προτύπων. Έπειτα μου έκαναν εντύπωση τα νούμερα που είπατε, όπως και στον κύριο Ντιπρέ, και μας μιλήσατε για την ανάγκη δημιουργίας σωστών αστυνομικών δομών σε χώρες της Βορείου Αφρικής κτλ. Και μας είπατε για τις καινούργιες ανάγκες σε προσωπικό, όμως πιστεύω πως ε, λίγα άτομα παραπάνω δεν θα καταφέρουν να επανθρώσουν την ε, αστυνομική επιτήρηση σε όλη τη Βόρεια Αφρική παρόμοιος και με την Ευρωπόλ. Πιστεύω πως οι τρεις ε, επιπλέον υπάλληλοι δεν θα τρομοκρατήσουν τους τρομοκράτες. Και γι' αυτό λοιπόν εντυπωσιάστηκα από το τι πιστεύετε πώς θα καταφέρουμε με λίγες θέσεις παραπάνω. Ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον προτείνεται τη συγχώνευση Ευρωπόλ και Σεπόλ. πολιτική επιστροφής τώρα από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ιδιαίτερα πιο μικρά κράτη-μέλη, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες να εφαρμόσουν σωστά την πολιτική επιστροφή. Ιδιαίτερα διότι δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν πόρους. Πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα πιο μικρά κράτη-μέλη έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει με ομαλό τρόπο. Χρειαζόμαστε επαφές και τη δημιουργία περισσότερων επαφών με αυτά τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να βοηθήσουμε. Η Σίλβη έχει το λόγο. Ήθελα να δώσω κάποια για τα οποία καλύφθηκα από τους προελίσσαντες συναδέλφους. Τέλος πάντων, ε, ωραία, πάρα πολύ θετικό όλα αυτά που μας είπατε. Αλλά θέλω να μου πείτε για κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή για αυτή την κατηγορία βοήθεια και το ε, πρόγραμμα της επανεγκατάστασης, είπατε για 25 εκατομμύρια, εάν δεν κάνω λάθος. Για πέστε μου, μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως ακριβώς συζητηθεί και για τα κράτη δικαιούχους. Ε, επίσης κάτι άλλο που δεν έχω καταλαβεί όπως και ο συνάδελφος Ντεπρέ. Αυτές οι θέσεις, αν κάνουμε μια απλή διαίρεση, αντιστοιχούν σε κάπου στα 33 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά, είναι για πλήρη απασχόληση. μας επίσης τι είδους θέσεις είναι αυτές. Ίσως είναι κάτι που να καταλάβει, δεν είναι απλώς για το πώς θα ε, καταπολεμήσουμε τα δίκτυα της διακίνησης στην ΙΑΙΖΟ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τώρα επόμενος. Είναι η κυρία Γκάλ, Κίνγκα Γκάλ. Κύριε Ρουέτα, για τη ΣΥΠΟΛ έχω αναλάβει κάποια έκθεση και προχωρήσαμε και στον τριμήρη διάλογο και κατάλαβα ότι ήδη είναι χρήσιμη υπηρεσία, θα είναι ακόμη πιο χρήσιμη για την μετανάστευση και είπαμε ότι προβλέπονται διάφορε δραστηριότητε εκπαίδευση, όλα αυτά θα τα διαχειριστεί η ΣΥΠΟΛ. Μήπω όμω θα πρέπει να προκοδοτήσουμε παραπάνω και αυτή την υπηρεσία, είναι σημαντικό. Ακόμα και αν αυτό δεν γίνει το 15, Α γίνει το 16. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ. Πιόρκα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, γενικώ έχω σκεφτεί ότι μετά τις τραγωδίες των οποίων γίναμε μάρτυρες, το μόνο που νιώθω είναι απογοήτευση. Γιατί αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς θα σταματήσουν τα ανθρώπινες ζωές και όσον αφορά τις διασώσεις δεν έχουμε κανένα κονδύλιο να προβλέπετε. Δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Μόνο για τη Frontex κουβεντιάζουμε. Δεν είναι σωστό. να συγκρίνουμε τις επιχειρήσεις της Frontex με το Mare Nostrum και να ε, αγνοούμε το τι γίνεται τη σημερινή μέρα. Και είναι θλιβερό ακριβώ το ότι τα κρατημέλη δεν κάνανε πολλά για να σταματήσουν ε, την απώλεια των ζών και ό,τι κάνανε τέλο πάντων δεν κάνετε τον προπολογισμό. Λέμε για Frontex, για Europol, για επιτήρηση, για σωματοφύλακες, όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το ότι έχουμε ε, outsourcing και υπεργολαβία σε τέτοιες υπηρεσίες. Και αντίθετα με τους άλλους που πήραν το λόγο, εγώ θέλω να σας πω ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους υπεργολαβία ανάθεση στις σε εξωτερικές υπηρεσίες της φύλαξης των συνόρων. Άρα γι' αυτό και διστάζω, έχω επιφυλάξει αυτόν τον προπολογισμό. Επίσης, ε, ε, έχω δύο-τρεις ερωτήσεις που ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Κάτι όσον αφορά τις επιστροφές. Ανησυχούμε πολύ ότι αυτές οι ταχείες επιστροφές θα πρέπει να ενισχυθούν, να στηριχτούν. Και αυτό είναι προβληματικό στην πολιτική μας. Θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση σε, σε, σε επίπεδο προπολογισμού τέλο πάντων και να δούμε κατά πόσον χρησιμοποιούνται καθόλου χρήματα κοινοτικά για τις επιχειρήσεις στα ελληνικά ύδατα. Τι γίνεται. Για τέτοιες αποστολές προβλέπονται χρήματα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, συγγνώμη, κάτι άλλο έκανα να απομιλήσω αλλά δεν σας και Κοιτούσα τι προβλέπει ο προϋπολογισμός όσον αφορά αυτή την διευρυμένη γεωγραφική περιοχή. Και θα αναρωτήσω ε, και ο ίδιος, τι θα πει διευρυμένη γεωγραφική περιοχή. Συμπάθατε με που δεν πρόσεχα λέγατε. Η τελευταία αγορητής, η κυρία Λόριστεν. Διευκρινίστε λίγο αν θέλετε. Τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση. Αφορά πολλά κράτη-μέλη. Τι προβλέπετε σαν ποσοστώσεις, σαν ε, προσαρμογή των ποσών, την αριθμική. Πώς ακριβώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα, πώς προβλέπετε να αξιοποιηθούν. Πώς θα υπάρξει έλεγχος τη αποτελεσματικότητας τη χρήση των πόρων. Πολύ σημαντικές ερωτήσεις και λεπτομέρειες. Άρα εδώ θα βάλουμε τελεία και θα ζητήσουμε να απαντήσει ο κύριος Γενικός. Ευχαριστώ, Κλώδη. Να σας πω για τον τριπλασιασμό τη προοικοδότησης ή τέλος πάντων τριπλασιασμό των επιχειρήσεων. Πρώτα πρώτα. Έχουμε αυτά τα 9 εκατομμύρια που κάπου περιφέρονται. Όμως άμα δείτε τις πραγματικές δαπάνε της Frontex για, για τον Τρίτονα και τι γίνεται από πλευράς Ιταλίας, καταλήγουμε στο να δαπανάτε διαφορετικό ποσό κάθε μήνα. Υπάρχει προγραμματισμό για το τι θα γίνει το καλοκαίρι, θα γίνει το χειμώνα. Δεν είναι επομένω ετησίω ούτε πάντα 3 εκατομμύρια, ούτε πάντα 9 εκατομμύρια. Αυτό να μην ξεχνάτε. Αν θέλετε τέλο πάντων να σα βρω τα στοιχεία. Από το 1 διακινείται μέχρι το 3. Οπότε, ανάπτυξη λοιπόν των όσων έχουμε, τον όσων έχουν τα κράτη-μέλη. Μια αγορά φτάνουμε στο 90%, αλλού λιγότερο το, το ποσοστό της κάλυψης και επίσης πόσες ώρες αφιερώνονται ε, και αυτό είναι με μεταβλητή και το κάνει πολύ μπερδεμένο. Άρα προσπαθούμε τώρα να κάνουμε αυτό το οποίο γίνεται και στα πλαίσια του Μαρενάστρου. Δηλαδή συνεργασία και ένταξη του συστήματος μας στη δράση των Ιταλικών αρχών και έχουμε αυτή την επέκταση της επιχειρηματικής ζώνης με το τρίτον. Έτσι θα συνεργαστεί η Frontex με την Ιταλία, θα κινητοποιηθεί ε, περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο υλικό, περισσότερος κόσμος. Όλα αυτά θα είναι στα πλαίσια της εντολής της ε, Frontex. Αλλά η αναζήτηση και η διάσωση γίνεται τώρα και η περιπολία, τέλο πάντων η επιτήρηση της επιχειρησιακή ζώνης μας δείχνει ότι υπάρχει κόσμος που χρειάζεται βοήθεια. Οπότε ακριβώς με το πρόγραμμά μας είπαμε ότι περισσότερο θα πηγαίνουμε τώρα από ό,τι στο παρελθόν με την ε, σωτηρία ε, των ανθρώπων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορώ να σας παράσχω αν θέλετε. και θα διαπιστώσετε ότι ακριβώς τριπλασιάζουμε τις επιχειρησιακές ενέργειες και εδώ έχουμε κάποια κρατημέλη τα οποία συμβάλλουν με δυνάμεις και αυτό το κάνουν δωρεάν δεν ζητούν κάλυψη πάρα πολύ σημαντικό αυτό Α, παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο αν όλα αυτά μένω τα λάβετε υπόψη πρέπει να σταθούμε περήφανοι ω Ευρωπαίοι που τελικά αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Και κάναμε μια πολύ σημαντική στροφή στην πολιτική μας. Δεν είναι τώρα ώρα να ξεκινήσουμε πολιτική κουβέντα, αλλά λάβετε υπόψη ότι του αμέσω επόμενους λίγους μήνες πρόκειται να γίνει μια συζήτηση όσον αφορά ε, την φύλαξη των συνόρων στα πλαίσια του θεματολογίου για την μετανάστευση. Και πιστεύω πραγματικά ότι και στο Κοινοβούλιο και στο ε, Συμβούλιο διαπιστώθηκε τον Απρίλιο ότι κάτι πολύ διαφορετικό ξεκίνησε και γεννήθηκε όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων. Κάτι πολύ διαφορετικό από το τι είχαμε μέχρι σήμερα. Έχουμε και κάποιε επιχειρήσει της ΚΕΠΑ, αλλά δεν καλύπτονται από τη δική μας προϋποδότηση. Ε, εμείς ε, έχουμε αναλάβει ε, έλεγχο από πολίτε, όχι από μέσα στρατιωτικά. Έχουμε ακτοφυλακή και έχουμε και κέντρα τα οποία τα διαχειρίζονται πολίτε. Άρα δεν υπάρχει κάποια σχέση βρικοδότησης τη Frontex με την ΚΕΠΑ. Τώρα για το θέμα της τρίτης χώρας που είπατε. Ναι, ναι, τα 7 εκατομμύρια όντω σταγόνα του ωκεανού. Όμω το πρόγραμμα μας εκεί τρέχει τώρα. Δηλαδή σε σχέση με περιφερειακή ανάπτυξη και προστασία. Οπότε κάπως βοηθάμε. Και βλέπουμε και μέσω του θεματολογίου ότι έτσι επαναπροσανατολίζουμε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Μας απασχολεί δηλαδή και όσον αφορά την ανάπτυξη ε, η μετανάστευση. Οπότε κινητοποιούμε ό,τι μπορούμε, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάπτυξης μόνο. Μιλάμε τώρα για κάποια περιορισμένη, περιορισμένο τομέα, όπου εκεί πέρα ενεργούμε. Εκεί είπαμε θα ρίξουμε 8 εκατομμύρια φέτος και άρα 7 εκατομμύρια θα τα προσθέσουμε τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά το πρόγραμμα περιφερειακής ε, ανάπτυξη και προστασία. Αλλά θα έχει συνέχεια αυτή η υπόθεση. Κύριε Ντεπρέ, πολύ σωστά τα είπατε. Θίξατε ακριβώς το πιο δύσκολο σημείο. Όπου το είπαν και άλλοι, ε, και η κυρία Χολμάγκερ και άλλοι συνάδελφοι, ότι κινούμεθα αναγκαστικά στα πλαίσια του ισχύοντος πλαισίου για τις θέσεις των υπαλλήλων. Τελικά θα υπάρξει μια καινούργια ανακατανομή. Όπως ξέρετε υπάρχει 1% περικοπή της υπηρεσίες, είναι 1% όπως και στην Επιτροπή που πάνε εκεί για την ανακατανομή, οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς θα μετακινήσουμε ε, ανθρώπινους σπόρους από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Αυτό γίνεται. Θα δείτε τον προπολογισμό τον οποίο συζητούμε και θα τον εγκρίνουμε την Τετάρτη για το 2016. Και όλο και κάτι θα προσθέσουμε για αυτές τις τρεις υπηρεσίες του 2016. Και για την κυρία Κίνγκελ που θέλω να πω ότι στο μέλλον θα διαπιστωθεί πόσο χρειάζεται η ΣΥΠΟΛ μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση και ο οργανισμός. Αν τι να κάνουμε, υπάρχει στενότητα δημοσιονομική. Ναι, η Άζο θα πρέπει σίγουρα να ενισχυθεί στο μέλλον. Είμαι εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτών των τριών υπηρεσιών και προς το παρόν προσπαθούμε να δούμε ε, τι θα γίνει φέτος μας, κανομένοι προς το παρόν. Υπάρχει το θέμα των προσλήψεων, να βρούμε δηλαδή ε, κόσμο γιατί για το άσο δεν είναι αυτό πάντα τόσο εύκολο. Μην ξεχνάτε πάντως ότι σε πολλές από αυτές μας τις κινήσεις κινητοποιούμε ανθρώπινους πόρους των κρατών μελών. Θα κάνουμε δηλαδή που δεν ε, καλύπτονται από αυτές τις θέσεις, όπως και με τη Frontex. Αυτή η 16, ε, για την Europol ας πούμε, τους έχουμε εκεί για να μας βοηθήσουν να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη που διαθέτουν ε, δυνάμεις και πόρους ε, για τις υπηρεσίες. Να γίνει διαχείριση των χρημάτων, να γίνει κάποιο συντονισμός. Και κοιτάξτε, είμαι συντηρητικός, ε, ολιγαρχής, δεν ζητάω πολλά και όσον αφορά τις ε, θέσεις. Um, uh, also to Madame Guillaume, uh, to certain extent, uh, Αυτά που λέω αφορούν και τα όσα ρώτησε η κυρία Guillaume. Ναι, ναι. Όντως πολλές αυτές τις θέσεις δεν είναι πλήρως ε, απασχόλησης. Ε, κάποιες από αυτές επίσης είναι αρκετά υψηλόβαθμοι πάλι γιατί αφορούν, ε, αφορούν την ε, διαχείριση. Τώρα, όσον αφορά τα χρηματικά ποσά αυτών των πόρων, θα δείτε για τη χρήση του 2016 ότι υπάρχουν πλέον πόροι για τις ε, επανα, επανεγκαταστάσεις. Κύριε Λόρεστεν, θα δείτε ότι στο θεματολόγιο προβλέπονται 50 εκατομμύρια. Υπάρχουν και οι πόροι επίσης για την επανεγκατάσταση στα πλαίσια του προγράμματος του Οπότε θα δείτε ότι όσον αφορά την κατάσταση. Ε, θα υπάρξει πιο θαραλέα πολιτική, πιο τολμηρή πολιτική από την Κομισιόν. Αυτά, Πρόεδρε, και όποιος θέλει, διμερός μπορούμε να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, συναδελφοί, διμερός. Επίσης, στη σημερινή συνάντηση των συντονιστών θα προσπαθήσουμε να αποφασίσουμε αν θα γνωμοδοτήσουμε και αν ναι θα ορίσουμε και η συντάκτη. Γιατί για μας είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήσεις σας και ευχαριστώ και σας για τις απαντήσεις. Θα συνεχίσουμε να προσέχουμε τα σημαντικά δημοσιονομικά θέματα. Τώρα, συνάδελφοι, περνάμε στην κατάσταση στη Μεσόγειο. Τις επόμενες δύο ώρες θα ασχοληθούμε με αυτό και παρακαλώ τους ομιλητές να έρθουν εδώ στο Προεδρείο ενώ εγώ θα σας εξηγώ τι θα κάνουμε τώρα. Συνάδελφοι, την περασμένη εβδομάδα θα μάθατε για τη δήλωση για τη μετανάστευση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Έγιναν πολλές αναφορές στα βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων διάσωσης και των εγκαταστάσεων των μεταναστών, αλλά πρέπει να αναλυθούν και οι λόγοι αυτών των μεταναστευτικών ροών και των απελπισμένων προσπαθειών ανθρώπων να περάσουν στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Σήμερα λοιπόν οι ομιλητές θα μιλήσουν συγκεκριμένα για αυτά τα στοιχεία Ιδιαίτερα η ανταλλαγή απόψεων θα επικεντρωθεί στο θέμα της στρατηγικής συνεργασίας με τρίτες χώρες και ιδιαίτερα για τα προγράμματα περιφερειακής προστασίας, επιστροφών και των λόγων της μεταναστευτικής αυτής ροής. Την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια έγιναν είπα οι δηλώσεις Συμβουλίου και Επιτροπής και έπειτα η διαχείριση των συνοριακών ελέγχων και ο Frontex και άλλων υπηρεσιών θα συζητηθούν. Στις δύο αυτές ώρες λοιπόν θα Έχουμε τους δύο τον Ρομπέρτο Μασούλα και τον κύριο Σίλκι Άγκε. Και θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα που σας ανέφερα. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητάς. Αν αποσιάζει κανείς να μας το πείτε. Πέτρο Σεράνο, που ασχολείται με την επιχειρησιακό συντονισμό από την εξωτερική, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Για πρώτη φορά μας έχουν στείλει ομιλητή. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Σεράνο. Μετά ο William Lacey Swing, Γενικός Διευθυντής του Διεθνής Οργάνωσης για τη Μετανάστευση. Μετά ο κύριος Μιχαήλ Άγχελ Μορατίνος, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας που ευγενώς δέχτηκε και μάλιστα σε πολύ γρήγορα να προσέλθει. Θα έρθει, θα έρθει σε λίγο. Έρχεται. Τέλος. θέλαμε να ακούσουμε τον καθηγητή Steve Pierce που πολύ τον ξέρετε από το Πανεπιστήμιο του Essex και τη νομική σχολή του αλλά δυστυχώς αρέστησε και παραμένει κλινίδης. Αυτοί είναι οι ομιλητές. Πρώτα οι εισηγητές όπως κάνουμε συνήθως. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συγκυρία για να γίνει αυτή η δεύτερη ανταλλαγή απόψε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Ροβέρτος Μασούλα και μετά η Σεσίλ Κέρνγκέι και μετά ο, ο Ρομπέρτο. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλωσορίζω και τα μέλη του πάνελ. Συναντώμαστε μετά τη νέα στρατηγική της Κομισιόν για τη Μετανάστευση κάτι το οποίο είναι θετικό και χαιρόμαστε για το ότι η Κομισιόν και η Κοινοβούλιο συμφωνούν σε πολλές προτάσεις και ιδιαίτερα στην ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης της μετανάστευσης η οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξωτερικές πτυχές. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί με το να κοιτάει η Ευρώπη μόνο στο εσωτερικό της είναι όλο και υψηλότερο τύχη. Πρέπει να δούμε πώς θα σώζουμε τους ανθρώπους στη θάλασσα και τι μέλλον θα έχουν στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να δούμε και παραπέρα και να αντιληφθούμε πως οι εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Ως πολιτικοί πρέπει να κοιτάμε πέρα από την πενταετία μας ε, και να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Και άρα πρέπει να επαναξετάσουμε και τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες, τις χώρες προέλευσης και να δούμε τις αιτίε του φαινομένου και το τι μπορεί να γίνει για να βοηθήσουμε τις χώρες ειδικά στην υποσαχάρια Αφρική για να σταθούν στα πόδια τους. Πρέπει να δούμε δηλαδή τους παράγοντες που εξωθούν τους ανθρώπους αν ε, δεν υπάρχει μέλλον στις χώρες τους θα φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί εξαρτήτως τι γίνεται και θα πεθαίνουν στην έρημο ή στις θάλασσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει την σχέση της με τρίτες χώρες, να δούμε πού πάει η ανθρωπιστική βοήθεια και το εάν χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Βεβαίω και τα δίκτυα των διακινητών πρέπει να καταπολεμηθούν, αλλά δεν μπορεί να είναι η αρχή και το τέλος της εξωτερικής διάστασης και εάν μπορούν να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη σε στρατιωτική δράση νομίζω πως θα πρέπει να συμφωνήσουν και στην αντιμετώπιση των άλλων πτυχών της μετανάστευσης. Θα πρέπει να έχουμε στοχευμένη βοήθεια στην συνοριακή πολιτική, στην βοήθεια στις τρίτες χώρες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις αιτίες του φαινομένου είναι μέσω της ε, οικοδόμησης δυνατοτήτων μακροπρόθεσμα. Και εδώ πέρα παίζετε εσείς τον σημαντικό ρόλο και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Επίσης στηρίζω την σύσταση ε, δυνατοτήτων ε, υποδοχής εκτός ε, της Ένωσης για να πληροφορούν για τις δυνατότητες νόμιμης εισόδου. Παραδείγματο χάρη για τους σκοπούς ε, σπουδών. Ένα μικρό αλλά απαραίτητο βήμα. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει για τον κόσμο πριν φτάσουν να μπουν σε σκάφη που δεν είναι αξιόπλοα ακούμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι ε, αναζητούν προστασία και τελικά τους λένε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα μέχρι να φτάσουν στην Ευρώπη και ουσιαστικά τους οθούν ε, στα χέρια των διακινητών. Η προσέγγιση της Ευρώπης πρέπει να βελτιωθεί και οπωσδήποτε εδώ πέρα υπάρχει η μεταγκατάσταση. Είδαμε πως η Κομισιόν ζητάει τη μεταγκατάσταση 20.000 ατόμων από θείας από τρίτες χώρες αρκεία. Ε, αυτός ο αριθμός. Τόσο είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Επίσης, σε συνεργασία με την υπηρεσία ασύλου, πρέπει να υπάρξουν κάποια κριτήρια για να είναι αποτελεσματική η μετεγκατάσταση, για να αυξήσουν τα κρατημέλη τις δυνατότητες υποδοχής και να βοηθήσουν στη γρήγορη ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων. Δεν αρκεί να μπουν σε ένα αεροπλάνο, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να ζήσουν. Όταν μιλάμε σε ανθρωπιστικές περιπτώσεις, τα νόμιμα μέσα για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε μέσα όπως ανθρωπιστικές βίζες, εκπαιδευτικές βίζες πρέπει να ε, τα εξετάσουμε. Γεγονό είναι πως η πόρη μας δεν είναι απεριόριστοι πρέπει όμως να διασφαλίσουμε πως οι περιορισμένοι αυτοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για αυτούς που αξίζουν προστασία. Όσοι δεν αξίζουν προστασία πρέπει να επιστραφούν. Ε, σεβόμενοι βεβαίως πλήρως στις αρχές της μη επαναπρόθεσης πρέπει να δούμε τις διαδικασίες επανεισδοχής με, τρεις, με χώρες και να εφαρμοστούν αυτές. Το φρούρι Ευρώπη δεν είναι η απάντηση αλλά είναι και το να μην έχουμε έλεγχο των συνόρων μας πρέπει τα κράτη να μπορούν να λειτουργούν αλλά όχι εις βάρος των ανθρωπιστικών μας υποχρεώσεων. Πρέπει λοιπόν να έχουν και οι δύο πτυχές τους απαραίτητους πόρους. Τώρα όσον αφορά την υπηρεσία ασύλου πρέπει να αναπτυχθεί για να γίνει ένα σημαντικός εταίρος των κρατών μελών στον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων όπως η πληροφόρηση, η επανεκατάσταση και η κατάρτιση. Εγώ ζητούσα και θα συνεχίσω να ζητάω η Άσο να κάνει περισσότερα και είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Η Άσο μπορεί επίσης να εγγυηθεί μια κοινή εποπτεία της εφαρμογής και των βέλτιστων πρακτικών. Οπότε αναμένω την σημερινή συζήτηση και γνωρίζω πως θα αντλήσουμε αρκετά διδάγματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι στη δήλωση του Συμβουλίου του την περασμένη εβδομάδα έγινε λόγος για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε με τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε τους λόγους της Cecil τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συζητητές που είναι εδώ αυτή την σημαντική στιγμή. Ξεκίνησε αυτή επομένως, η πολιτική διαδρομή, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να γίνει μια στροφή στην προσέγγιση προ τη μετανάστευση πλευρά τη Ευρώπη, γιατί από αυτό το φαινόμενο δεν καταπολεμείται, αλλά ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, σε όλη του τη σφαιρικότητα και στο σύνολό του. Άρα χρειάζονται κάποια ε, μέσα βραχυπρόθεσμα επίγοντος χαρακτήρα, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να περιμηθούμε αυτές τις αξίες που δεν θα τη ζωή. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια διάσωση για αυτές τις βασικές αξίες και να μην έχουμε αυτές τις στήρες πολεμικές των κρατών μελών που έχουν προκλητικό χαρακτήρα. Οπότε ε, ακόμα δεν έχουμε καμία ε, απάντηση, τίποτα που να βλέπουμε μακριά, αλλά αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι μια ριζική διαφορά στην ε, δραστηριοτική πολιτική και να μπορέσουμε έτσι μακροπρόθεσμα κάτι να κάνουμε. Όχι στο υποστατικό, αλλά στο διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο. Άρα έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι βαθιέ ρίζε του φαινομένου τη μετανάστευση και επίση θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην διεθνή σκηνή και πώ θα εμπλακούν όλοι τα κράτη-μέλη, διεθνείς οργανισμοί, κοινωνία των πολιτών και οι τρίτες χώρες. Όλοι θα πρέπει να συνεργαστούν για μια ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικά κοινή όσον αφορά τη μετάφραση. Επίση, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε κάθε πολιτική, κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μα, ούτω ώστε να έχουμε τον καλύτερο συνδυασμό εσωτερική και εξωτερική πολιτική και κυρίω θα πρέπει να κατευθύνουμε την αναπτυξιακή μα πολιτική σε κάποιε συγκεκριμένε ε, λύσει ε, και αυτό αναφορά την φτώχεια, την ασφάλεια, τις διώξεις που αυτές είναι οι βασικές αιτίες της ε, παράτυπης μετανάστευσης που αναγκάζει τον κόσμο να μεταναστεύσει. Και είδαμε το πώς, μάλλον να δούμε πώς δεν θα ε, κάνουμε κάτι εκ των υστέρων και στο τέλος της διαδρομής, αλλά πολύ πιο νωρίς όσον αφορά αυτού του είδους τη μεταξύ αυτά τα κύματα μετανάστευσης που τελικά μόνο το τέλος τους ε, αντιμετωπίζουμε. Άρα θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση ε, της μετανάστευσης, να έχουν προγράμματα ε, μετεγκατάστασης ή μάλλον επανεγκατάστασης και θα πρέπει με αυτούς οι οποίοι συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια να υποστηρίξουμε περισσότερο μια μεταναστευτική πολιτική ε, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με αλληλεγγύη και με το να μοιραστούμε τις ε, ευθύνες και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το 85% των προσφύγων ζουν στο Νότο και στην Ευρώπη και στις ε, αναπτυγμένες χώρες είναι μόλις το 14% γιατί μιλούμε για άλλο μισό εκατομμύριο που έρχονται ε, στις βιομηχανικές χώρες αλλά περιμένουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις γιατί αν δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη κανένα κράτος μέλος από μόνο του δεν μπορεί να βοηθήσει για το φαινόμενο αυτό το οποίο από την ε, φύση του ε, είναι συνεχές, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Είναι κατακλείδη, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την επανεγκατάσταση αλλά και την μετεγκατάσταση. Αυτό τώρα μας απασχολεί και σίγουρα να δούμε και πώς θα μπορέσουμε αυτές τις προτάσεις να προωθηθούν και κάποια κρατημέλη τελικά να δεχθούν ε, και τα άτομα από Ερυθρέα αλλά και από τη Συρία. Είναι κάτι το οποίο αφορά πολλές χώρες οι οποίες έχουν ε, κινητοποιηθεί. Ε, δεν είναι μόνο αυτές οι δύο χώρες, είναι πολύ περισσότερες. Άρα έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και ε, τη ίσως για αυτήν την ε, πολύ καλή εισαγωγή και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σεράνο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία σας βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής μας, ιδιαίτερα για να σχολιάσει τις δηλώσεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τα πρόσφατα γεγονότα στη Μεσόγειο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να δώσετε έμφαση ιδιαίτερα στα όσα συνέβησαν στην Μεσόγειο και να προσπαθήσετε να αναλύσετε τις θέσεις σας παρά να μας παρουσιάσετε απλά το γενικό πλαίσιο της δράσης της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να εστιάσετε στα συγκεκριμένα ζητήματα, να αναφερθείτε στη Λιβύη και στις εταιρικές σχέσεις με, και τις συνεργασίες με τις τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ, τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και μάλιστα σε ένα πάνελ με τόσο διακεκριμένους προσκεκλημένους όπως τον κύριο Σουίν. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται, έχει την ίδια άποψη με την Ευρωπαϊκή, με το, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντική αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουν προκύψει με τις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπίσουμε τα αίτια του φαινομένου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση είναι πανέτοιμη να τα αντιμετωπίσει. Επίσης χρειάζεται φυσικά μια ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, και ακριβώς αυτό πιστεύουμε στην Υπηρεσία Εξωτερικής δράση. Και πράγματι, ένα από τα πλεονεκτήματα των ε, όσων θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια των εργασιών μας ε, είναι αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία λοιπόν πλαισίου διμερών και πολυμερών ε, σχέσεων που θα στηριχτεί φυσικά οικονομικά οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως Υπάρχει επίγουσα ανάγκη λόγω των εξελίξεων στη Μεσόγειο, λόγω των πιέσεων από πολλά κράτη-μέλη και φυσικά λόγω των ε, πολυαριθμών θανάτων αυτών των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να σταματήσει και είναι κάτι που δεν γίνεται να ανεχτούμε. Να σας πω επίσης ότι οι συγκρούσεις που έχουν οξύνει την κρίση είναι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν και άλλες επιπτώσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Στην παρουσίασή μου θα επικεντρωθώ σε αυτά που ζητήσατε κύριε Πρόεδρε. Έχω χωρίσει σε τέσσερα σημεία την παρουσίαση. Καταρχάς νότια γειτονία, τι κάνουμε με τις γειτονικές μας χώρες, επίσης το πλαίσιο συνεργασίας, το τι κάνουμε στις χώρες ε, διαμετακόμισης και τέλος πώς αντιμετωπίζουμε τις ε, ένοπλες συγκρούσεις. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, να σας πω ότι είναι πανέτοιμη να αναλάβει το συντονιστικό αυτόν ρόλο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική διάσταση της ε, ατζέντα της στα πλαίσια του δικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει συνεργασία ε, ανάμεσα στην Προεδρία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην υπηρεσία μας έτσι ώστε ο συντονισμός να είναι όσο το δυνατόν καλύτερος. Ένα από τα βήματα που ήδη έχουν υλοποιηθεί και είναι κάτι οριζόντιο είναι ο διάλογος με τις ε, σημαντικότερες χώρες. Εκεί θα στείλουμε συνδέσμους για θέματα μετανάστευσης στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Και επίσης, να σας πω ότι η μετανάστευση είναι μόνο ένας από τους πυλώνες του προγράμματος. Υπάρχουν και άλλα μέσα στα πλαίσια αυτά. Είναι ο διάλογος, η κινητικότητα, η ασφάλεια, οι συνεργασίες κινητικότητας για παράδειγμα, η διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνιών ε, υποδοχής μαζί φυσικά με οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την μετανάστευση και την κινητικότητα, αποτελούν ένα κομμάτι της πολιτικής μας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της κινητικότητας και η ανάγκη αντιμετώπισης ε, του φαινομένου των σχέσεων των γειτονικών μας χωρών με τις δικές τους γειτονικές χώρες. Επίσης, ενίσχυση ε, σχέσεων με το Μαρόκο, την Τινησία και την Ιορδανία. Έχει δημιουργηθεί ε, διάλογος με το Λίβανο και έχουμε αρχίσει διαδικασίες για έναρξη διαλόγου με την Αίγυπτο για θέματα κινητικότητας και μετανάστευσης γίνονται διαπραγματεύσεις για διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων. Αυτό να σας πω είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα και χρειάζεται πολύ προσεκτική αντιμετώπιση από όλες τις πλευρές. Επίσης ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις με την Τινησία για το ίδιο θέμα. Ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος έχει μεταβεί στις περιοχές αυτές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και επίση να σας πω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εκδόθηκαν πρόσφατα, η Τουρκία αναδείχθηκε σε έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στην περιοχή αυτή. Υπάρχει μια συμφωνία υποδοχής που ετέθησε ισχύ τον Οκτώβριο του 2014 Γίνεται διάλογος αυτή τη στιγμή για την διευκόλυνση ε, των, ε, της έκδοσης θεωρήσεων και τη διευκόλυνση των ε, ταξιδιωτών από την Τουρκία. Φυσικά ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ε, Τουρκία, ιδιαίτερα στα σύνορά της, διότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχει δεχτεί η χώρα 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία. Η υπηρεσία μας, λοιπόν, θέτει την Τουρκία ως ε, κύρια προτεραιότητα Θέλουμε να παρέχουμε συνδρομή και συνεργασία και επίσης ε, αυτό θα το πραγματοποιήσουμε μέσω της αποστολής ε, κάποιου συνδέσμου από την ε, Frontex. Επίσης το πλαίσιο συνεργασίας για κινητικότητα και μετανάστευση στη Μεσόγειο και Αφρική. Θα ήθελα να τονίσω ότι το γενικότερο πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα σε Ευρώπη και Αφρική για μετανάστευση και κινητικότητα περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης και πολιτικές δηλώσεις. Τον Απρίλιο του 2014 στην Σύνοδο Κορυφής εγκρίθηκαν κάποιες ε, αποφάσεις οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο πακέτο για τη μετανάστευση και το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε την συνέχιση του διαλόγου και την χορήγηση κονδυλίων. Επίσης, σε διαδικασία του Ραμπάτ και του Χαρτούμ. Η διαδικασία του Ραμπάτ άρχισε το 2006 στο Ραμπάτ, συγκεντρώνει 55 χώρες Ευρώπης και Αφρικής, κυρίως από την Βόρεια Δυτική και Ανατολική Αφρική. Επίσης, το Νοέμβριο του 2014 είχαμε την ε, δήλωση της ε, Ρώμης με τις ε, προτεραιότητες που συνδέουν τη μετανάστευση και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των εγκλημάτων που συνδέονται με αυτή. Τον Ιούνιο θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας, θα επικεντρωθούμε περισσότερο στη χρηματοδότηση των διαφόρων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων ταμείων. Επίσης, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ε, εντοπίσουμε το κύριο πρόγραμμα το οποίο θα συντονίσει τα υπόλοιπα, θα επιτρέψει η ανταλλαγή πληροφοριών για την ε, αποτροπή της ε, παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος. Αυτές είναι οι κυριότερες εξελίξεις Καλύπτουμε επίσης την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τις χώρες του ε, κέρατος της Αφρικής. Ο διάλογος αυτός άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο στη Ρώμη. Πρώτη συνεδρίαση της ε, Συντονιστικής Επιτροπής τον Απρίλιο. Στο πρώτο στάδιο εξετάζεται η διακίνηση ανθρώπων και η συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου ανάμεσα στο κέρας της Αφρικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, υπάρχει και η διαδικασία της Βουδαπέστης, λιγότερο σχετική με, ε, το θέμα μας, η οποία βέβαια ασχολείται με, την, με τις σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία. Να σας διακόψω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη. Και με αυτό εννοώ αυτήν την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση και μπορεί να σας ε, φαίνεται κάπως ε, ήπια η διατύπωση, όμως ε, πιστέψαμε δεν είναι καθόλου. Είχαμε και μία δήλωση την περασμένη εβδομάδα σχετικά με αυτές τις ε, συνεργασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς θα κληθείτε να απαντήσετε σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα τόσο δύσκολα ζητήματα, τους διακινητές, για παράδειγμα, είναι πραγματικά δύσκολα σημεία για συζήτηση και μπορούμε να συζητούμε όσο θέλουμε. Όμως τώρα έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Υπάρχουν συγκρούσεις στη Λιβύη, συγκρούσεις στη Συρία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επικεντρωθείτε σε αυτό και στο πώς η υπηρεσία εξωτερικής δράσης βλέπει την κατάσταση στη Συρία και τη Λιβύη. Είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν τώρα και θα μας ρωτήσουν τι κάνουμε. Ποια λοιπόν είναι η δική σας ε, ανάλυση και προοπτική. Αυτές είναι ερωτήσεις τις οποίες ε, κάνουμε και για τις οποίες θέλουμε πιστεύω όλοι απαντήσεις. Συνεχίστε. Θα προσπαθήσω να αλλάξω κατεύθυνση. Όχι, δεν ήθελα να σας φοβήσω. Αλλά να μιλήσετε και γι' αυτό γιατί αυτό είναι το θέμα που μας ενδιαφέρει. Καλά. Βέβαια οι σειράξεις είναι σημαντικό τμήμα της ανάλυσης μας. Ελπίζω να μην αναμένετε καμία μαγική λύση από μένα. Όχι, κοιτάξτε, αυτά είναι δικαιοδοσίες του Συμβουλίου. Αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε και από εσάς. Κοιτάξτε, εδώ βασικά πρέπει να συνδυάσουμε τρία στοιχεία. Την πολιτική διαδικασία ή μάλλον, ή μάλλον έτσι μια γενικότερη θεώρηση των σειράξεων που έχουμε μπροστά μας. Ναι, ναι, όχι, συνεχίστε, συνεχίστε. Μάλιστα. Κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι σειράξεις αυτές έχουν συνδιασυνδεόμενη δυναμική μεταξύ τους. Είδαμε πως η σύραξη στη Συρία προχώρησε και στο Ιράκ κατά κάποιον τρόπο και στην Ιεμένη. Υπάρχει ένα περιφερειακό πρόβλημα στη Μέση Ανατολή το οποίο δηλητηριάζει την κατάσταση και στη Μεσόγειο και στη Λιβύη και επίσης δηλητηριάζει την κατάσταση στη Σομαλία γιατί μπορεί να υπάρξουν μεταναστευτικές ροές από την Ιεμένη στη Σομαλία κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια περιφερειακή σύραξη και δημιουργείται μια νέα ισορροπία δυνάμεων. Επίσης υπάρχει μια θρησκευτική διαμάχη. Αυτό είναι το μείγμα που αντιμετωπίζουμε. Αμείς τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε. Προσπαθώ να μιλήσω made a statement, we know that, and you know, we, we, you know, we're supportive of what she has to do. συνδέονται όλα αυτά με την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Να μας πείτε δηλαδή ποια είναι τα δυσκολότερα στοιχεία για σας. Ας πούμε στην πράξη πώς θα αντιμετωπίσετε τους δουλεμπόρους ή τι θα γίνει με τις εταιρικές ε, συμβάσεις σε περιπτώσεις ε, εμφυλίου ας πούμε αφού μιλάμε για εταιρικέ σχέσεις εντάξει όταν είναι σταθερή η κατάσταση όταν όμως είναι ασταθής αφού μιλάμε για επανακατάσταση Συρίων ή Σύρων σε άλλες χώρες πώς τα βλέπει αυτά η ΕΔΑ την περασμένη εβδομάδα μας είπανε ορισμένα πράγματα. Εσείς πώς τα βλέπετε από την πλευρά της ΙΕΔ, τις εταιρικές σχέσεις. Ξέρουμε τι γίνεται στη Συρία και τη Λιβύη, δεν ξέρουμε όμως ποια είναι η δική σας προοπτική της ΙΕΔ, πώς να στο πω. Της ΙΕΔ. Κοιτάξτε, άλλα κάνουμε σε άλλες χώρες. Η Συρία είναι η πιο δύσκολη χώρα. Αλλά τι κάνουμε, τι κάνουμε στη Συρία. Να σας πω τι κάνουμε στη Συρία. Να σας πω. Αν μου λέτε ότι το ξέρετε. Όχι, ξέρουμε τι κάνετε από τη δήλωση. Τέλος πάντων, συνεχίστε, συνεχίστε. Τι προσπαθούμε να κάνουμε στη Συρία. Είναι να σταθεροποιήσουμε την πολιτική διαδικασία. Αλλά δεν στοχεύεται αυτό βλέπω. Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την πολιτική διαδικασία, προσπαθούμε να στηρίξουμε μόλις υπάρξει ο κατάλληλος χώρος στη Συρία μια λειτουργούσα δημόσια διοίκηση που να μην για να μπορέσει να δημιουργηθεί σωστή διακυβέρνηση στη Συρία governance προσπαθούμε να στηρίξουμε τις εξελίξεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Συρία και προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις της ριζοσπαστικοποίησης στη Συρία. The Syria, uh... Βέβαια δεν είναι μεμονωμένη η σύραξη στη Συρία, είναι τμήμα της γενικότερης περιφερειακής κατάστασης και πρέπει να συνεννοηθούμε με τους, με όλους τους παράγοντες όπως στη Σαουδική Αραβία είναι κυρίως διπλωματική προσπάθεια ναι, διπλωματική σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία την Τουρκία, το Ιράν ένα από αυτά που κάνει διπλωματικά η Ένωση για να αλλάξει η δυναμική στην περιοχή είναι η στήριξή μας για τις ε, συνεννοήσεις για τα πυρηνικά του Ιράν ας πούμε. Αυτά είναι σαφή στοιχεία, σαφή. Κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος φυσικά όλοι γνωρίζετε, όλοι γνωρίζετε ότι μία από τις προτάσεις από τα στοιχεία που πρότεινε το Συμβούλιο ήταν ε, να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα στη Μεσόγειο προφανώς και αυτό θα σήμαινε ότι χρειάζεται η στήριξη και των χωρών της περιοχής. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με αυτές. Αν τεθούν συγκεκριμένα ερωτήματα με τα χαράς να τα απαντήσω, αλλά η διαδικασία και ο σχεδιασμός συνεχίζεται και επίσης διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία μια ενός νομικού υποβάθρου ετοιμάζεται ένα ψήφισμα και από το Συμβούλιο Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη τεχνικές λεπτομέρειες τώρα συγκεκριμένη συνεργασία με συγκεκριμένες χώρες αυτά είναι θέμα εσωτερικών Υπουργείων Εσωτερικών όχι η ΕΔ οι τοπικές οργανώσεις ασφαλείας δηλαδή κτλ. Εμείς ε, είμαστε το γενικότερο πλαίσιο για να το πω έτσι, το γενικότερο Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Τι είναι τώρα. Κοιτάξτε, μην μιλάτε σε μένα στην Επιτροπή. Α, στην Επιτροπή, ναι, στην Επιτροπή. Ξέρουμε ότι έχετε διπλωματικές δραστηριότητες και παίζετε διπλωματικό ρόλο. Όλα τα ξέρουμε στην Επιτροπή μας. Αλλά να σας επαναλάβω χωρίς να σας ενοχλήσω. Η εξωτερική υπηρεσία θα ήθελα να μας πείτε πολύ συγκεκριμένα τι κάνει. Έχουμε τη Συρία, έχουμε τη Λιβύη και δημιουργούν και οι δύο χώρες πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν απέναντι στη Μεσόγειο και συζητήσαμε πολύ και τα, το, το δουλεμπόριο, μας τα είπε και η κυρία Μογκερίνη την προηγούμενη εβδομάδα, μία προοπτική να μας δώσετε από πλευρά της ΙΕΔ. Μερικά αναπάντητα ερωτήματα, δηλαδή τι κάνει το Συμβούλιο ή θα κάνει ας πούμε για αυτά που είπατε για τις εταιρικές σχέσεις. που σχετίζονται και με τη δική σας δουλειά. Αυτό θέλω να ακούσουν πολλοί συνάδελφοι. Γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Τι γίνεται με τα πλοία, τι γίνεται με τις επιστροφές. Πρακτικά πράγματα δηλαδή. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Συνήθως δεν παρεμβαίνω έτσι, αλλά, αλλά να. Να, αυτά ήθελα να σας πω και να μας πείτε. Λυπάμαι που δεν ανταποκρίνομαι σε αυτά που θέλετε ή που αναμένατε. Πολλά από τα ερωτήματα ως προς το πώς γίνονται οι επιχειρήσεις στη Μεσόγειο ή θα γίνουν ακόμη συζητιούνται συζητιούνται με τους διάφορους παράγοντες και ό,τι κάνουμε θα γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο με σεβασμό των δικαιωμάτων όλων εκείνων που, εμπλέκονται και τους αιτητές ασύλου και, ασύλου και τους μετανάστες αλλά όλα αυτά τα ξέρετε είπατε, τα ξέρετε, μάλιστα. Καλά, δεν αναμέναμε να παραβιάσετε το διεθνές δίκαιο, εντάξει. Υπάρχει κανένα άλλο βασικό στοιχείο που θέλετε να μας πείτε. Αν ναι, πέστε τα. Ίσως το τελευταίο. Οι άλλες επιχειρήσεις ΚΠΑ ναι, όχι τα, τα, πες τα. Μα αφού τα ξέρετε όλα. Ε, δεν πειράζει, πέστε τα ξανά. Μήπως απλώς να μου θέσετε ερωτήματα. Εμένα ο ρόλος μου είναι απλώς συντονιστικός και ελπίζω να ξέρετε ποιες είναι οι αδυναμίες και ενός συντονιστού στις επιχειρήσεις ΚΠΑ μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Κοιτάξτε, η ανταπόκριση και ο συντονισμός, η κρίση και ο είναι κάτι γνωστό. Εμείς μιλάμε για την κρίση στη Μεσόγειο, αυτό θέλουμε να είναι, η Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο. Μα το είπα, το είπα, είπα ότι προσπαθούμε να λύσουμε τις πολιτικές διαδικασίες που επισυμβαίνουν εκεί, που είναι πολύπλοκες, πολύπλοκες. Αλλά και αυτό το ξέρετε και επίσης προσπαθούμε να στηρίξουμε τις χώρες που είναι στη δεύτερη γραμμή για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των το Μαλί, τον Νίγηρα για να αυξηθούν οι δυνατότητες ασφάλειας αυτών των χωρών και ένα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ήταν να ενδυναμωθεί η επιχείρηση στον ήγυρα ίσως με αποστολή προσωπικού και υπάρχει και ένα σχέδιο μαζί με το IOM για ένα κέντρο συντονισμού ή πληροφόρησης στον Νίγηρα και στον Νίγηρα για να ασχοληθεί ακόμη και με θέματα επανεγκατάστασης προσφύγων. Αυτό είναι όμως πειραματικό πρόγραμμα. Θα δούμε πού θα πάει και μέχρι πού μπορούμε να κινηθούμε. Έχουμε επιχείρηση και στην ανατολική ακτή της Αφρικής. Ξέρετε ότι πολλοί προέρχονται μετανάστες από εκεί, από την Ερυθρέα, τη Σομαλία, το Σουδάν. Αλλά έχουμε επιχειρήσεις εκεί. Τη δημιουργία, ας πούμε, κράτους στη Σομαλία. Κράτους για διασφάλιση και διοργάνωση των ε, αστυνομικών και στρατιωτικών της δυνάμεων, δυνατότητες θαλάσσιας προστασίας, αυτά ε, κάνουμε εκεί. Και επίσης με, ασχολούμαστε με τις πολιτικές διαδικασίες, η υπάτη εκπρόσωπος είναι σε επαφή με τον Περναρδίνο Δελεόν, αλλά και ιδίω για τη συνέχεια. Τι θα γίνει εάν όπως ελπίζουμε υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη. Πρέπει μετά να μπορούμε να διαθέσουμε πόρους για να στηριχτεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που θα δημιουργηθεί ώστε να υπάρχει ασφάλεια στα βασικά τουλάχιστον. Να αυτά είναι αυτά με μεγάλη φρόνηση η οποία όμως δεν έχει τελειώσει ο σχεδιασμός της. Τώρα για τη UNAFOR, όπως σας είπα, μόλις ελήφθη η απόφαση και προφανώς θα πρέπει μετά να υπάρξουν σαφείς κανόνες για το πώς και πότε και πού θα εναποθέσουμε ανθρώπους που θα έχουμε σώσει από κίνδυνο θανάτου αλλά δεν μπορώ να σας τα πω πιο συγκεκριμένα δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό ακόμα συζητιέται από τα κράτη-μέλη, δεν έχει συμφωνηθεί. Αλλά θα υπάρξει απόφαση, καθώς και το τι να κάνουμε με τους δουλεμπόρους. Ξέρετε τι κάναμε με τη Σομαλία, στη Σομαλία, αλλά αφού ακόμα συζητιέται δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Μπορούμε να έχουμε διάφορες υποθέσεις και σενάρια, και ε, θα ήθελα να σας ακούσω αλλά δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Θα πρέπει να γίνει η συμφωνία και, και συντονισμός αλλά δεν έχει ακόμα γίνει. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ήδη νομίζω έκανα κατάχρηση του χρόνου σας. Αν έχετε ερωτήσεις να απαντήσω. Ναι, θα υπάρξουν νομίζω ερωτήσεις. Σας κατευχαριστούμε. Και τώρα πάμε τον κύριο Λέισε Σουίνγκ. Γενικό Γραμματέα του Διεθνού Οργανισμού για τη Μετανάστευση, που βεβαίω και έχει εμπλακεί σε όλα αυτά τα θέματα. Ευτυχώ που ήρθατε εδώ και παρακαλώ έχετε τον λόγο. Κύριε Πάτρα. κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, είναι για τον οργανισμό μας μια τιμή το να ανταλλάσσουμε σήμερα απόψεις για μια σφαιρική, ολοκληρωμένη πολιτική μεταναστεύση που είναι κάτι που χρειάζεται και που όλοι να θα αποκτήσουμε. Θα ήθελα να σα πω ότι για μα είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το θεματολόγιο τη Ένωση. Είναι μια ε, πρωτοβουλία, είναι ένα πρώτο βήμα ε, σε μια αρκετά μακρά διαδρομή. Επίσης, πιο συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ θετικό το ότι η ψήφιση προτεραιότητά σα είναι να σώσετε ανθρώπινε ζωέ. Είναι μια θέση που ανέκαθεν ε, την προωθούσαμε γιατί αν σώσετε τι ανθρώπινε ζωέ, τότε υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ ε, για του λογικού. Έχουμε επομένω μια παλιά δέσμευση για να προχωρήσουμε σε μια σφαιρική πολιτική. Και θέση μας ανέκαθεν ήταν ότι η μετανάστευση είναι αναπόφευκτη και για δημογραφικού και για άλλου λόγου. Οπότε και αυτό το οποίο χρειάζεται απολύτω είναι να έχουμε τι δεξιότητε που χρειάζεται. Αν θέλουμε να έχουμε τι δουλειέ που χρειάζεται για να πάνε, πάνε καλά οι οικονομίε μα. Δεν ξέρω ποιε είναι ε, ε, οι, προγνώσει, αλλά λένε ότι χρειάζεται περίπου 40 εκατομμύρια παραμονεργαζόμενα για τα μέσα του αιώνα. Οπότε και μέσα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχουν εργατικά χέρια, αλλά πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχε πολιτικές, πολιτικές ανθρώπινες και υπεύθυνε. Γι' αυτό και εγώ θέλω να σας αναπτύξω ποια είναι τα παράδοξα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ίσως δεν μπορούμε να τα άρουμε, θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Και Ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλούμε για ένα μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Πάμε στην Παγκόκ, την Παρασκευή. Περιφερειακή διάσκεψη θα γίνει εκεί για τους μετανάστες στην Βενγκάλη και στη θάλασσα του Άνταμαν. Οπότε αυτό που ήθελα να σας αναπτύξω είναι το ότι δεν είναι πρόβλημα προς επίλυση μετανάστευση. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει κανείς να την διαχειριστεί και αν δεν την διαχειριστεί τότε ε, η μετανάστευση θα διαχειριστεί εμάς. Τα τρία θέματα, τα εξής θέλω να σας πω πρώτα-πρώτα. Η Μεσόγειος στο μέσον της τέλειας καταιγίδας. Για να δούμε στην παγκόσμια σκηνή, σαν πλαίσιο τι γίνεται. Χρειάζονται λόγια και περισσότερο. Μιλάμε για ένα δίσανα, εφτά Και έχουμε πάρα πολλούς που για πρώτη φορά αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Όπω λένε τα στατιστικά, έχουμε πάνω από 50 εκατομμύρια τώρα. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ρεκόρ. Επίση, είναι χώρες προηγούμενο αυτές οι τρομερές συγκρούσεις, οι πόλεμοι που γίνονται ταυτόχρονα και δημιουργούν ανθρωπιστικές κρίσεις. Από τη Δυτική Αφρική μέχρι την Ασία. Και δεν υπάρχουν και τόσε πολλές οάσεις ενδιάμεσα όπως το θέλαμε. Και επίσης τώρα δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια διαδικασία, κάποια μέθοδος πολιτική βιώσιμη ή κάποιο διαπραγμάτευση που να τρέχει τώρα και να δίνει κάποιε ελπίδε για μέσω βραχυπρόθεσμη λύση. Ελπίζω, προσεύχομαι να βγω λάθο. Επίση, χωρίς προηγούμενο, σε αυτή την ε, περίοδο έχουμε ε, πάρα πολλά αισθήματα κατ' μεταναστών, σχεδόν ε, ξενόφοβα και νομίζω ότι έχουμε όλο ένα και λιγότερη εμπιστοσύνη του κόσμου στις δυνατότητες που έχουν οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις να διαχειριστούν την μετανάστευση με κάποιο τρόπο λογικό. Τέλος, υπάρχει κενό ηγεσία. Λείπει το πολιτικό κουράγιο και θάρρος. Και επίσης δεν υπάρχει ηθική νοημοποίηση. Ολόνα και συρρυκνώνεται όσον αφορά το ότι ολόνα και πιο συχνά παραβιάζεται το Γι' αυτό και μιλώ για την τέλεια ε, καταιγίδα που μας περιβάλλει. Και θεωρούμε και αισιόδοξου, φανταστείτε. Αλλά εγώ έτσι θα το έλεγα, ότι εκεί βρίσκεται η Μεσόγειος. Αν θέλουμε για να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις βράχη μέσω μακροπρόθεσμες και επίσης για να δούμε ποιες είναι οι αιτίες της μετανάστευσης. Είναι τέτοιες που η μετανάστευση μεγάλης κλίμακας θα παραμείνει χαρακτηριστικό φαινόμενο του αιώνα μας. Πάλι, μακάρι να βγω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω. Μιλάμε για δημογραφικά αίτια, μιλάμε για τον γεράσκοντα βορρά, μιλάμε για θέσεις απασχόλησης που ε, υπάρχουν κενές και επομένως ε, συνέχεια πολλοί και περισσότερο μεταναστεύουν, γι' αυτό κάναμε και το του γιατί από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Νοέμβριο έχει σωστό άνθρωπο ζωή. Και έχουν με περίπου 2.000 μετανάστε οι οποίοι πνίγηκαν στην Μεσόγειο χωρί το Στρομή. Ε, αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα και γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι τώρα το έχει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα. Επίσης έχουμε και αυτές τις τραγωδίες, έχουμε την ε, ψηφιακή παράδοση όμως. Ε, πάνω από το 1 τρίτο ε, του κόσμου σε όλη την υδρόγειο είναι συνδεδεμένη, ίντερνετ. Και άλλοι παράγοντες υπάρχουν. Ζήτηση εργατικών χεριών. Και οι οικονομικές διαφορές βορρά-νότου κλπ. Άλλο θέμα τώρα. Τι θα κάνουμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το στρατηγικό πλαίσιο, συνεργαστήκαμε μέχρι τώρα. Κατέβασαμε τις ιδέες μας μετά την ε, τραγωδία της Λαμπεντούσα τον 8 του 2013 και είχαμε αυτά τα 368 φέρετρα στην αμμουδιά της Λαμπεντούσα. Ε, αυτό μας έπεισε ότι πρέπει να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Όλες αυτές τις προτάσεις λοιπόν. Και ο καθένας έχει τις, τα δικά του σημειώματα, τις δικές του προτάσεις, αλλά τελικά συγκλίνουν. Το λέμε παγκόσμιο αποτύπωμα. Το λέμε ευκαιρία να βοηθήσουμε. Τι θα πρέπει να κάνει κανεί. Πρώτα πρώτα, να σώσει ανθρώπινε ζωέ. Να σεβαστεί τα δικαιώματα των μεταναστών. Δεύτερον, να εντοπίσει τι αιτίε του φαινομένου για την παράνομη μετανάστευση. Ναι. Με ασφάλεια επομένω και αξιοπρέπεια να υπάρχει κινητικότητα του κόσμου αυτό το υποσώστοση που προτάθηκε ε, είναι κάτι θετικό, αλλά θα πρέπει να αυξηθεί, θα πρέπει να ανέβει. Ξέρω ότι διαφωνούν τα κράτη-μέλη, αλλά είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να γίνουν κι άλλα. Έχουμε τώρα 16,7 εκατομμύρια μετανάστες. Έχουμε εκτοπισμένους 30 τόσα εκατομμύρια που όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται και έχουμε εκτοπισμένους μέσα στη Συρία όσους έχουμε και εκτός Συρίας. Αλλά θα πρέπει τώρα να δούμε τι θα γίνει με τις θεωρίες διαβατηρίων τις ανθρωπιστικές. Το πώς θα έχουμε ανθρωπιστική διαχείριση των συνόρων. Και οι τέσσερις γείτονες της Συρίας, οι έξι της Λιβύης δεν νομίζω ότι ποτέ έλαβαν κάποιο, κάποιο είδου ευχαριστώ και του αναγνώρισε από το αυτό που κάνει γιατί συνέχεια ε, με μεγάλο τίμημα έχουν έρθει τα σύνορα. Ένα εκατομμύριο έχουν μπει στην φτωχή Ιορδανία. 200.000 χτες, ε, πέρσι ε, πήγανε ε, στον Λίβανο επίσης που είχαμε 5 εκατομμύρια πληθυσμό και υπεστήριξε ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες. Επομένως, θα πρέπει να γίνει τέτοιος διαχείριση των σύνορων. Θα πρέπει τα σύνορα να θεωρηθούν στοιχείο ανθρωπιστικό. Κυκλική μετανάστευση και ρύθμιση των θεωρήσεων, ε, μεταγκατάσταση, όλα αυτά που ξέρετε πολύ καλά. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία του χαρτιπορίου που θα μας βοηθήσει να τα πάμε καλύτερα από ό,τι είπαμε στο παρελθόν. είναι στόχο του να υπάρξει κάποιο είδου εταιρική σχέση, όπω θα είπε ο κύριος Σεράνο, διάλογοι που έχει ενεργοποιήσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην με γρηγορούμε, αλλά τελευταίο θέλω να αναφέρω αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι οι προκλήσεις. Τρεις είναι αυτές οι προκλήσεις. Ε, είναι και θεωρητικό και πολιτικό χαρακτήρα και πρέπει επομένω αυτέ τι προκλήσει να τι αντιμετωπίσουμε. Αλλιώ θα αποτύχουμε τελικά. Πρώτη πρόκληση. Να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε το αφήγημα το σχετικό με την ε, μετανάστευση που τώρα είναι δηλητηριώδες. Και σας διαβεβαιώ γιατί η χώρα η δική μου έτσι οικοδομήθηκε. Με τα χέρια, με τις καρδιές των μεταναστών. Οπότε όλα ήταν θετικά σαν πνεύμα, σαν αφήγημα. Ε, εκεί θα πρέπει να επανέλθουμε, σε τέτοια σοβία. Κανεί δεν λέει ότι είναι άγγελοι οι μετανάστε. Μα δεν είναι καν οι συμπατριώτε μα. Ε, άγγελοι όλοι. Όμω θα πρέπει τώρα να έχουμε ένα τέτοιο πνεύμα που να μην είναι δηλητηριώδε και να υπάρχει περισσότερη ισορροπία και να καταλήγουμε στο ότι η μετανάστευση όσο αφορά την ανάπτυξη είναι πάντοτε χρήσιμη. Πάνε χέρι-χέρι μετανάστευση και ανάπτυξη πέρα από τα στερεότυπα. Ποια είναι ότι έρχονται να πάρουν τις δουλειές μας. Ε, Φέρνουν αρρώστιες, είναι εγκληματίες και τώρα μετά το Σαρλί Εμπδο είναι και τρομοκράτες. Μα δεν έρχονται με αυτά τα σκάφη των ε, δουλεμπόρων. Ε, οι τρομοκράτες έχουν άλλους τρόπους. Οπότε αυτά τα, αυτές τις ιδέες θα πρέπει να διαχειριστούμε, ώστε να σταματήσει αυτή η μυθολογία και το στίγμα προς τους μετανάστες. Άλλη τώρα ε, πρόκληση που έχει σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τη διαφορετικότητα. Δεν ξέρω πώς με αυτές τις αιτίες που σας είπα, κυρίως τις δημοκρατικές αιτίες, δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε χωρίς να αλλάξουμε βαθιά τις κοινωνίες μας. Νομίζω ότι το Έθνο κράτου του 19ου αλλάζει, αλλάζει τρόπο στα μάτια μας. Θα πρέπει να γίνουμε πιο πολυεθνικοί, πιο πολυπολιτισμικοί. Με πολλές ε, θρησκείες ταυτόχρονα που μας υπάρχουν αν θέλουμε να πετύχουμε για αυτούς τους στόχους. Και για να πετύχουμε χρειάζεται πολιτικό θάρρος, χρειάζεται επένδυση. Ενημέρωση του κόσμου. Παιδεία, εκπαίδευση. Συνειδητοποίηση με εκστρατείες για το τι γίνεται με τη μετανάστευση και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μεταναστεύουν και επίση θα πρέπει να μετακινηθεί η συζήτηση από το θέμα τη ταυτότητα στο θέμα των αξιών. Μόφα κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια για την Βρετανία. Είναι Βρετανός, δεν είναι Σομαλός. Μιλά σαν και εμένα. Και τελικά σημαίνει τι ίδιε αξίε. Αυτό είναι η μετανάστευση. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Αυτό το οποίο ε, λέω, το πώς θα συγκεράσουμε το παράδοξο της, το να υπάρχει ταυτόχρονα εθνική κυριαρχία και ταυτόχρονα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Αυτά θα πρέπει να συγκεράσουμε. Εθνική ασφάλεια και ανθρώπινη ασφάλεια. Και κατακλείδη κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση θα πρέπει να βαδίσουμε. Είμαστε ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς όσα έκανε για τα βήματα πρόοδου που κατάφερε. Έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο μπροστά μας, αλλά κάναμε καλή αρχή. Και εμείς θα σας ε, στηρίξουμε και εμείς και οι άλλοι εταίρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον κύριο Μορατίνο, στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας. Καλώς ήρθατε. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τις απόψεις σας πάνω στο θέμα. για δέκα λεπτάκια, γιατί ξέρω πως οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και όπως είπε και ο κύριος Λέισι Σουίνγκ αυτό θα είναι το πιο καλό κομμάτι της συζήτησης. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε και πρέπει να σας πω πως είναι μεγάλη μου τιμή που επανέρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καλό να έρχεται κανείς ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό συμφώνησα αμέσω ε, στην συμμετοχή μου σε αυτό το πάνελ γιατί νομίζω πως όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούμε να μοιραστούμε τις ευθύνες ε, που είχαμε στο παρελθόν. Και η προηγούμενη ισπανική κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει κάποιες παρόμοιες στιγμές παράνομης μετανάστευσης ε, το έτος 2000, από το 2006 μέχρι το 2010 και επικεφαλής ε, της ισπανικής διπλωματίας ε, ήμουν εγώ και προσπαθούσα να βρω τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Οπότε Παρά το ότι αναγκάστηκα να ξυπνήσω 5 ώρα το πρωί από το Λονδίνο, να πάρω τρένο και ταξί για να έρθω εδώ πέρα, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον ύπατο πρόσωπο και την ομάδα του γιατί νομίζω πως επιτέλους, επιτέλους κατάφερε να βάλει το θέμα της μετανάστευσης ε, ε, επιτάπτως και στην κορυφή της ατζέντας και να ευχαριστήσω και τις δύο συνεισηγήτριες ε, τις κυρίες Μέτσολα και Κιέγγε για την ε, συνάντηση αυτή πάρα πολύ επίκαιρη. Ευχαριστώ τον είπα το εκπρόσωπο, τον Πέτρο Σεράνο και τους συναντήφους για τη δουλειά που έκαναν, αλλά όπως ε, είπε ο φίλος μου εδώ πέρα είναι το πρώτο βήμα εδώ πέρα λοιπόν... Έχετε θέσει τη μετανάστευση στο κέντρο, γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο και αναφέρθηκαν οι συνεισηγήτριες στις αιτίες της μετανάστευσης, αλλά να πω, Πέτρο, με κάθε σοβαρότητα πως τα μέτρα που έχετε εγκρίνει είναι απολύτως απαραίτητα σε όλους τους τομείς, ασφάλεις, ασφάλεια, εμπλοκή κτλ. Όλα αυτά, από όλα αυτά λείπει μία λέξη, η διπλωματία. Για τον λόγο αυτό θα πω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου της ε, Ισπανικής ε, κυβέρνησης στις Κανάριες νήσους, στη Ούδα και Μελίγια κάθε μέρα μπαίνανε 2-3 χιλιάδες άνθρωποι και υπήρχε τρομερή ε, πίεση όπως σήμερα οι Ιταλοί φίλοι μας. Τι κάναμε λοιπόν. Οργανωθήκαμε κάθε Παρασκευή πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με όλους τους υπουργούς εσωτερικών, οικονομικών, εξωτερικών, η υπηρεσία πληροφοριών κάθε Παρασκευή για να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε την κατάσταση. Και όλοι είχαν κάτι συγκεκριμένο να κάνουν. και μετά λέγαμε τι θα κάνουμε. Η πρώτη απάντηση ήταν πάμε στην Ευρώπη να ζητήσουμε από τους Ευρωπαίους να μας βοηθήσουν. Και πήγαμε στην Κομισιόν, στην Υπατή Εκπρόσωπο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μας δίνανε απαντήσεις ε, έτσι ήξης αφήξης ε, δεν απασχολούσε το θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση ναι εντάξει φέραμε τη Frontex αλλά ε, η Frontex δεν μπορούσε να κάνει όσα περιμέναμε. Οπότε πρέπει, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε διμερή διπλωματία. Γιατί ερχόταν στην Ισπανία. Εντάξει, η Ισπανία ανθούσε και τα λοιπά, αλλά ήταν και στα σύνορα της Ευρώπης και ερχόταν από την Αφρική και την Ασία. Τα πλοία και οι βάρκες που πήγαιναν στα Κανάρια ήταν γεμάτες ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές, τον Νεπάλ, από όλο τον κόσμο. Διέσχιζαν την Αφρική, πήγαιναν στη Γάμβια, Γουινέα, Κονακρή, μετά Κανάριες νήσους και καμιά φορά στην Αλγερία και το Μαρόκο. Οπότε αποφασίσαμε να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάποιες επισκέψεις, ε, να αλλάξουμε την διπλωματία μας. Εγκρίναμε ένα σχέδιο για την Αφρική, τριπλασιάσαμε την βοήθειά μας ε, στην αναπτυξιακή, στην Αφρική. ακούσαμε ε, ούτε μία λέξη για αναπτυξιακή βοήθεια στην Ήπειρο. Θα μου πείτε ότι σήμερα η κατάσταση διαφέρει. Ναι, συμφωνώ, γιατί έρχονται από τη Συρία, τη Λιβύη, λόγω των συγκρούσεων. Εγώ θα ήθελα τα πραγματικά νούμερα σήμερα. Το ένα είναι ότι η Λιβύη ε, δεν ελέγχεται και βεβαίως υπάρχει αυτή η αναρχία. Αλλά για τα νούμερα τώρα δεν ξέρω, βλέπω κάτι εικόνες στην τηλεόραση και έχω κάποιες πληροφορίες ότι ο κόσμος από την Υποσαχάρη Αφρική, την Ασία, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Και ομολογώ εδώ πέρα την άγνοιά μου, αλλά θα πω πως τουλάχιστον το πολύ 30% να είναι από τη Συρία και τη Λιβύη και άλλες συγκρούσεις τα υπόλοιπα 70% και πάνω είναι από την υποσαχάρια Αφρική γιατί πεινάνε. Δεν έχουν δουλειές, αξιοπρέπεια κτλ. Αυτές είναι οι αιτίες. Κύριε Μέτσολα, κύριε Κίνγκ, αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς για τον λόγο αυτό. Εγώ μεταφέρω, στους, λέω στους φίλους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνετε άμεση διπλωματία, όχι μέσω μη επανδρομένων αεροσκαφών. Πηγαίνετε στις χώρες. Μιλήστε με τους αξιωματούχους. Δεν ξέρω αν έχει... υπήρξε μια επίσημη επίσκεψη για τη μεταναστευτική πολιτική. Εγώ πήγα πέντε φορές στην Αφρική, άνοιξα τέσσερις ε, ε, πρεσβείες, ε, τριπλασίασα τον προϋπολογισμό μου για κατάρτιση, για απασχόληση, για την εκπαίδευση του κόσμου, πώς να ψαρεύει στη Σενεγάλη, στη Γάμπια. Κάτι έπρεπε να γίνει. Ξέρω τι κάνετε στον Νίγηρα και στο Μαλί. Αλλά αγαπητέ μου φίλε Πέδρο, μιλάς, μιλάτε για ανάπτυξη στρατιωτικών. Νομίζετε πως μόνο με στρατό και πολιτική ασφαλείας θα ε, λύσετε αυτά τα προβλήματα ο αγαπητό μα φίλος εδώ πέρα λέει πως αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο, κύριο Σουίνγκ, κάθε χρόνο, κάθε κάτι. Όχι, πρέπει να αλλάξει η πολιτική της Ένωσης για την περιοχή και οι Αφρικανοί είναι έτοιμοι, αυτό περιμένουν. Ζητάμε μια, ε, ζητήσαμε μια ευρωαραβική σύνοδο στο Ραμπάτ ε, και πήγαμε τελικά καλέσαμε όλες τις αφρικανικές χώρες και αποκαλέσαμε τη άσκηση ανάπτυξη και μετανάστευση γιατί χρειάζεται ανάπτυξη για να έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να δουλέψει εκεί πέρα αυτό πρέπει να γίνει και είχαμε μια μικρή επιτυχία ως ισπανική κυβέρνηση από 5.000 άτομα που ερχόταν κάθε μέρα στα Κανάρια να έχουμε μηδέν αφήξεις το 2009-2010. Μηδέν. Και όχι μόνο λόγω της κρίσης. Γιατί έχουμε συνεργασία με την Σενεγάλη, τη Γάμπια, το Μαρόκο και άλλες χώρες. Και ε, ψάχναμε ένα κοινό πρόγραμμα. Αυτό χρειάζεται λοιπόν. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Συμφωνήσαμε νομίζω και, και η Επιτροπή και οι Υπουργοί Εσωτερικών κάνουν καλή δουλειά, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Είναι η δουλειά τους ε, και λένε ότι δεν τους θέλουμε στα σύνορα. Μα ωραία, τότε πρέπει να σκηθεί η εξωτερική πολιτική λοιπόν. Δεν είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής και εσωτερικών. Μπορεί να γίνει. Και πρέπει να το δούμε ανθρωπιστικά. Αλλά όσον αφορά τη στρατηγική της Ένωσης, είναι κυρίως ένα ζήτημα εξωτερικό. Και γι' αυτό χαίρομαι που το συζητάνε και οι συνάδελφοί σας στην Επιτροπή Εξωτερικών για την πολιτική μετανάστευσης. Και τέλος για να λυθεί το πρόβλημα. Μία αρχή υπάρχει. σε συνθήκες ε, όπως ε, της Λισαβόνας. Αλληλεγγύη, φίλοι μου. Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρώπης με άλλες χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί πραγματικά θέλουν όλοι να λάβουν το λόγο. Έχουν ζητήσει λοιπόν όλοι το λόγο και θέλω να ακουστούν όλοι. Εγώ θέλω να δούμε λοιπόν πόσο σχετικά είναι όλα αυτά με την τωρινή κρίση και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν. Όπως είπα λοιπόν, ακόμα και ο κύριος Κέρκοπ ε, έχει ζητήσει το λόγο. Όλοι άπαντες. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε ε, είναι το εξής. Θα λάβουν το λόγο όσοι τον ζήτησαν με σειρά προτεραιότητας. Και θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι για να καταφέρουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Θα μας πάρει ώρα λοιπόν, να είστε σύντομοι. Αρχίζουμε καταρχάς με τις εισηγήτριες. Η κυρία Ματσόλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη, γιατί θέλω να δώσω το λόγο και στους άλλους. Έχω τρία σύντομα σχόλια. Χαίρομαι πολύ που αναφέρθηκε το θέμα της διπλωματίας από τον κύριο Μωρατίνο. Ε, δούλεψε για την ε, κυβέρνηση της Μάλτας πολλά χρόνια και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όταν μια κυβέρνηση ασχολείται άμεσα με την χώρα προέλευσης των μεταναστών έχει καλά αποτελέσματα. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται από τους πόρους που υπάρχουν και από το πόσοι έρχονται από την χώρα προέλευσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Μάλτα είναι η Λιβύη. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διπλωματική συνεργασία. Όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι προσπάθειές μας δεν επαρκούν. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε, πιστεύω, να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της κυβέρνησης ε, στη Λιβύη. πρωτού αρχίσουμε να συζητούμε για επιστροφή στη Λιβύη ή για ανάληψη ευθυνών από την κυβέρνηση της Λιβύης. Φυσικά τα πλοία αυτά δεν έρχονται μόνο από την Λιβύη και όλοι όσοι φτάνουν από τη Λιβύη δεν προσπαθούν να δραπετεύσουν, να ξεφύγουν από την κατάσταση. Υπάρχουν και άλλοι. Τώρα κύριε Σουίν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση μία συνέντευξή σας στο BBC, στο CNN, δεν θυμάμαι, πριν από μερικές εβδομάδες την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα, που μας είπατε ότι η μετανάστευση είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να διαχειριστούμε και όχι ένα πρόβλημα πως επίλυση. Αυτό πιστεύω πως πραγματικά ε, συνοψίζει όλη τη δουλειά που κάνω εγώ και η συνεισηγήτριά μου και όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα φύγει το πρόβλημα, δεν θα λυθεί. Πρέπει να το διαχειριστούμε και μάλιστα με αλληλεγγύη. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στη συνθήκη και όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει να εισαχθεί η λέξη αλληλεγγύη στη συνθήκη. Και πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η αρχή της αλληλεγγύης να εφαρμόζεται κιόλα. Όχι μόνο να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα διακινητών, αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα σωθούν ζωές. Κύριε Μορατίνο, θα μας ενδιέφερε να μάθουμε για τις ε, διαρθρωτικές διαφορές ανάμεσα σε Λιβύη και Συρία, όταν θα έρθει η ώρα σας να απαντήσετε. Μάλιστα δεδομένου ότι δεν έχουν στην ουσία λειτουργικές κυβερνήσεις. Η κυρία Κέγγι έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τους εισηγητάς για την ε, βοήθειά τους, για την εισφορά τους. Και στην πρώτη μου ερώτηση θέλω να απευθύνω στον κύριο Σεράνο για να καταλάβουμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτού του, του Συμβουλίου Κορυφής της Μάλτας. Ποια είναι τα βασικά μέρη. Γιατί ε, να δούμε και ποιοι θα συμμετάσχουν. Κάτι άλλο θες και κύριο Σεράνο. Όντως θα πρέπει να καταλάβουμε τις ε, αιτίες του φαινομένου. Γιατί είναι επίσης και όλα αυτά τα άλλα, τα σημεία των συγκρούσεων και των ε, πολέμων, τα καυτά. Άρα θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, όπως είπατε, για αυτό το θέμα. Και τι προβλέπετε ως συγκεκριμένες λύσεις για αυτά τα καυτά σημεία, ας πούμε, για την, για την ε, Συρία. Δεύτερη ερώτηση. Για τον κύριο Λέισι Σουίν, για την Ερυθρέα. Είναι δυνατόν η προστασία ή όλα αυτά τα προγράμματα ή όσον αφορά την επανακατάσταση και μετεγκατάσταση όλα αυτά μπορεί να υλοποιηθούν για δύο εθνότητες δηλαδή για Σύρους και κατοίκους της Ερυθρέας τέλος πάντων αυτούς πρόκειται την Ερυθρέα και να δούμε τι γίνεται με αυτούς αλλά και τους άλλους πέραν αυτών των δύο κατηγοριών. Τι γίνεται όσον αφορά επίση τι αντιπροσωπή τη κοινότητα σε αυτέ τι χώρε, τι προβλέπετε. Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλ. Η Σεσίλια Βίξτρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς σήμερα που ήρθατε εδώ και επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι αναγνωρίστε την προσπάθεια των ε, θεσμικών οργάνων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε την μετανάστευση και όχι να την αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα. Αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Σχετικά με το μέλλον της Frontex, θα ήθελα να ακούσω περισσότερα, γιατί αυτή τη στιγμή η Frontex εγείται αποστολών διάσωσης, εντοπισμού και διάσωσης και ορισμένα κράτη-μέλη επιφορτίζονται περισσότερο με την, τις αποστολές αυτές. Η δική μου ομάδα, η ομάδα Άλντε, πιστεύει πως χρειάζεται αναθεώρηση ο κανονισμός για τη Frontex έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική η συνεισφορά από όλα τα κράτη-μέλη και επίσης ζητά μια αύξηση του προϋπολογισμού της καθώς και μια κοινοτική προσέγγιση στις ε, αρμοδιότητες της Frontex και στις ε, ενέργειες διάσωσης. Επίσης, επιθυμούμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ε, λιμενικού με κατάρτιση, ευρωπαϊκή κατάρτιση που θα προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εσείς τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να αλλάξει η οδηγία έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά και τι ασφαλιστικές δικλείδες πιστεύετε πως χρειάζονται για να προστατεύονται τα δικαιώματα των μεταναστών και διάφορων ευπαθών ομάδων, όπως για παράδειγμα θύματα διακίνησης, ανήλικη κτλ. Επίσης, χρειάζεται να συζητήσουμε για το πώς θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τις τρίτες χώρες και πώς θα λαμβάνουμε και θα αποστέλουμε και σχετικά με τις λεπτομέρειες της ε, παράτυπης μετανάστευσης, ίσως θα, ήταν καλό να προσπαθούσαμε να καταρτήσουμε όσους ήδη έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μη νόμιμα, έτσι ώστε να ενημερώσουν τους υπόλοιπους που σκοπεύουν να το κάνουν και τους κινδύνους που διατρέχουν. Ε, κύριε Λέισι Σουίνγκ, πιστεύω πως αναφέρατε ορθώς την κύρια αιτία, τη ρίζα του προβλήματος, όχι της μετανάστευσης, αλλά της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Και πιστεύω πως πολύ σωστά αναφερθήκατε σε αυτήν την ξενοφοβία και τη μυσαλλοδοξία που υπάρχει, το ρατσισμό ακόμα σε πολλά κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτή την έλλειψη ηγεσία που αναφέρατε, πώς την κρίνεται και τι προτείνεται για το επόμενο στάδιο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η έλλειψη ηγεσία που υπάρχει. Και επίσης, κάτι που πιστεύω ενδιαφέρει πολλούς από εμάς, η συνεργασία με τις τρίτες χώρες όπως ανέφερε και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ακούσει πολλές προτάσεις μέχρι τώρα. Εγώ όμως πιστεύω πως ως Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα πρέπει να αναθέτουμε σε τρίτους και στην προκειμένη σε γειτονικές χώρες τις δικές μας αρμοδιότητες. Για το άσυλο για παράδειγμα. Και αυτό δεν συμπεριληφθήκε στην ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως έχει συζητηθεί στα πλαίσια διαλόγων από πολλούς εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίση σε πολλά επίσημα έγγραφα πριν από την επίσημη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες που εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανάγκη. Και Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία, αυτές είναι οι χώρες που αντιμετωπίζουν αυξημένες εισρώες μεταναστών και όχι η Ευρώπη. Και επίσης χρειάζεται φυσικά ο διάλογος με τις άλλες χώρες, όμως πιο σημαντική είναι η σωστή και εύρυθμη συνεργασία, ιδιαίτερα με τις χώρες από τις οποίες φεύγουν. Και θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τις απόψεις σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, προσκεκλημένους. Ιδιαίτερα ε, τον κύριο Μαρτίνο. Με ενδιαφέραν πάρα πολύ αυτά που είπατε και όντως υπάρχει ένα θέμα με τις χώρες διαμετακόμισης. Ε, κύριε Σεράνο, αναφέρατε και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, η οποία δεν είναι ακόμα λειτουργική. Δεν έχει αναλάβει λοιπόν στην ουσία καθήκοντα, όμως η τραγωδία υπάρχει και συνεχίζεται και αυξάνεται. Τι γίνεται λοιπόν εκεί στη Δυτική Λιβύη. Η Δυτική Λιβύη ελέγχεται από την κυβέρνηση της Τρίπολης η οποία δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα και δεν υπάρχει επιθυμία από την, ε, με, ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις να συνεργαστούν για να καταπολεμήσουν τους ε, διακινητές. Και κάτι άλλο αναφέρθηκε σήμερα η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου για τη δημιουργία μιας κοινή στρατιωτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα οι παράγραφοι 7 και 8 αναφέρουν ότι αυτή η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει διάφορα, διάφορα πλοία και θαλάσσιες επιχειρήσεις στα χωρικά του ΣΥΔΑΤΑ και θα μπορέσει για παράδειγμα να θέσει επί την ε, κυριαρχία της τα σκάφη άλλων χωρών. Κύρια Φεράρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια ερώτηση προς τον κύριο Σερένα όσον αφορά είναι τον απολογισμό των μαγμάτων ε, και το πόρους που επιτίθενται. Δεν είναι σαφές. Οπότε μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικές με εκείνους τους ε, πόρους. δηλαδή πόσα ξοδεύουμε στις ιδιωτικές χώρες για το άσυλο πόσα για τη μετανάστευση, πόσα για όλα τα επιμέρους θέματα που έχουν σχέση με την μετανάστευση, με τους συνοριοφύλακες κλπ. Και ακριβώ στο βωμό της διαφάνειας θα έπρεπε να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε τέτοια ε, δεδομένα. Αυτό θα ήταν μια καλή πρακτική. Τώρα, να επανέλθω στην Euroform, ε, την επιχείρηση εκείνη. Το είπαμε και στην Ολομέλεια και ο ίδιος και ε, ο ίδιος έχει ασχοληθεί για το πώς θα ε, έχουμε περισσότερη ενημέρωση και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ε, ακόμα βέβαια βρίσκεται να εξελίξει κατάσταση, αλλά συγκεκριμένα πράγματα δεν μπορούμε να μάθουμε. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι μαθαίνουμε από τις εφημερίδες ότι οι επιχειρήσεις αυτές εκτίλησονται σε τρεις φάσεις συλλογή πληροφοριών και περιπολία, ε, κατόπιν παρακολούθηση και καταστροφή στη συνέχεια αυτών των ε, σκαφών. Και εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, δηλαδή κινείστε με άξονα αυτές τις τρεις φάσεις. Πεςτε μου επίσης, προτίθεστε να καταπολέμησετε με αυτόν τον τρόπο το οργανωμένο έγκλημα που αφορά ε, το δουλεμπόριο από ό,τι γνωρίζουμε, η πρόσβαση σε αυτά τα σκάφη είναι μόνο η τελική πράξη. Γιατί πάρα πολύ καιρό οι μετανάστες υφίστανται βία μεταχείριση αλλά και βασανιστήρια. Οπότε όλα αυτά τα οποία κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αφορούν πολλούς μήνες πριν την επίβασή τους στα σκάφη των διακινητών. Άρα εσείς τι κάνετε τώρα, πώς συνεργάζεστε από αυτού με τρίτες χώρες. Επίσης, για πέστε μου τι γίνεται με τη διαδικασία του χαρτούμ. Ακόμη, δεν έχουμε μάθει αρκετά και υπάρχουν πολλές αμφιβολίες. Ε, και τι γίνεται, συνεργασία με δικτατορίες, πώς έτσι εξασφαλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα κάτι τελευταίο σαν παράδοξο έχουμε αυτή τη συμφωνία την Γάλλο-Γερμανική, ούτως ώστε να υπάρχει το 2025 ναι να μην παθρωμένο σκάφο, ούτω ώστε να προβαίνει σε επιχειρήσει αναγνώριση και ελέγχου και να καταπολεμηθεί έτσι το οργανωμένο έγκλημα. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε, Ισκά. Ναι, πολλοί ρώτησαν για την επιχείρηση της ΚΠΑ. Θα ήθελα να μου πείτε μερικά ακόμα. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το θέμα για συνεργασία, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Δεν μας είπατε όμως τίποτα γι' αυτό. Πώς γίνεται η εποπτεία ή θα γίνει και συνδέεται με τα ντρόν που κυκλοφορούν στο Μαρόκο κλπ. Μήπως σκοπεύετε να δημιουργήσετε μία βάση λειτουργίας ντρόν στη Βόρεια Αφρική. Δεν είδα πολύ αυτοκριτική. Γιατί είναι γνωστό ότι οι σχέσεις της Ένωσης με τον Καντάφη δεν ήταν ακριβώς τέλειες ούτε και για αυτό το θέμα της αντιμετώπισης των μεταναστών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα προφανώς έχουν παραβιαστεί στη Λιβύη και κρατούνταν πολλοί κόσμο σε απαράδεκτες συνθήκες λοιπά Αλλά παρόλα αυτά η Ένωση έδινε αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς το βλέπετε και αυτό και για τον κύριο Σεράνο. Τώρα οι ρίζες της μετανάστευσης αυτού του είδους η Ένωση ίσως συνεισφέρει, συμβάλλει και αυτή δημιουργία τέτοιων λόγων μετανάστευση με το εμπορικά της προγράμματα, την αλληλευτική πολιτική κτλ. Γίνεται συζήτηση στην Κομισιόν μήπως πρέπει να αλλάξουν αυτά τα προγράμματα ώστε να μην καθίστανται οι φτωχοί φτωχότεροι στις τρίτες χώρες και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν όπως στη Δυτική Αφρική διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνθήκη όπου λέει ότι όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να καθοδηγούνται από την αρχή της απάλληψης της φτώχειας. Αυτό πώς εφαρμόζεται. Επίσης αναφέρθηκε η Ερυθρέα και θα ήθελα να γνωρίζω πώς συνεννοείστε με, τους, με την κυβέρνηση της Ερυθρέας για να σταματήσει η μετανάστευση και από εκεί. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτή η έξοδος. Πώς το χειρίζεστε αυτό αφού καλέσατε την Ερυθρέα στη διάσκεψη στη Μάλτα. Δεν ξέρω πώς θέλει να συνεργαστεί η Ένωση με την Ερυθρέα για να σταματήσει η μετανάστευση από εκεί. Κύριε συμφωνώ βασικά με όσα είπατε, αλλά δεν γνωρίζω πώς μπορεί η Ένωση ή και μονομενα τα κράτη-μέλη να δώσουν λύση με τις ποσοστώσεις και με τις επαναγκαταστάσεις των προσφύγων. Εδώ ίσως υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικής ηγεσίας που αναφέρατε κι εσείς. Ευχαριστώ. Η Γιώτομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις μου είναι σύντομες. Στον κύριο Σιρανό. Σεράνο. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε κάποιες ε, πληροφορίες για τη συμφωνία επανεισδοχής με την ε, Τουρκία. Ε, ήταν και στην εντολή της προηγούμενης Κομισιόν. Μετά αναφέρατε τις διαπραγματεύσεις με τη, Λιβύα, με τη Λιβύη. Είναι δύσκολο βεβαίως να διαπραγματευτεί κανείς όταν δεν υπάρχει συνομιλητής, αλλά ο υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης είπε πριν από λίγες μέρες ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα για να βοηθήσει τη Λιβύη με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και η Λιβύη δεν μπορεί να είναι εξωτερικό σύνορο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μας. Πολλές ερωτήσεις έγιναν από, την, από τις κυρίες Φεράρα και Κέλλερα αλλά σημαντικό είναι να πούμε αυτό το οποίο είπε και ο Ισπανός Μας διαφεύγει η σχέση μεταξύ ε, ειρήνης και ανάπτυξης ε, και μετανάστευσης και δεν υπάρχει αυτό στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και είναι ντροπή. Αντί να σώσουμε λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο στόχο έχει να κρατάει τον κόσμο έξω και τώρα αναπτύσσεται. Απλά λέω πω εάν δεν κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις ε, με σωστή βάση θα καταλήξουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι για το 2015 και δεν θα είναι αξιοπρεπές. Ανησυχώ πάρα πολύ για την στρατιωτικοποίηση, αναφέρθηκε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε τις προκλήσεις αυτές με όπλα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, λέμε πως θα δράσουμε. Λέει εδώ πέρα πως πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες ασφαλείας στον Ήχυρα. Συγκεκριμένα δηλαδή, τι θα γίνει εκεί, πώς καταπολεμάμε τις διακινητές. εμένα μου φαίνεται μια στρατιωτική αντίδραση σε κάτι το οποίο δεν είναι στρατιωτικό. Και νομίζω πως καλό είναι αυτό το οποίο υπόθηκε. Πόσο κοστίζουν αυτά τα πράγματα. ποιε είναι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού. Και τέλος μου φαίνεται πως ε, θα κανιβαλίσουμε τα χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας για να κρατήσουμε εκτός τους ε, πρόσφυγες ε, και μετανάστες. Για το Χαρτούμ τώρα και την Ερυθρέα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με δικτατορία για να μην φεύγει ο κόσμος από τη χώρα. Και θα ήθελα να ξέρω κάτι άλλο. Λέμε πως θέλουμε να καταπολεμήσουμε τους διακινητές, αλλά έχουν μία αγορά γιατί δεν δίνουμε νόμιμες διόδους για προστασία στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης πως κάποιες χώρες ε, ε, ταυτοποιούνται διάφοροι διακινητές, αλλά δεν είναι διακινητές. Είναι κάποιοι σε μια βάρκα που κρατάνε το τιμόνι και αφού πρέπει να κατηγορήσουμε κάποιον, συλλαμβάνονται άνθρωποι που δεν είναι διακινητές. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κίνδυνοι και με αυτή την προσέγγιση και ελπίζω να μην υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση στα λιβικά ύδατα. Ευχαριστώ κύριε μου. Ευχαριστώ σύντομη θα είμαι. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση γιατί μας επιτρέπει να κάνουμε και μία αρχή γεωπολιτικής ανάλυσης. Νομίζω ότι πρέπει τελικά να χαρούμε για τη σύνδεση που γίνεται μεταξύ αυτής της γεωπολιτικής και των μεταναστευτικών ρόλων. Τρία θέματα θα ήθελα να θέσω, αν και μερικά θα έχουν θέσει άλλοι. Το πρώτο, τα προγράμματα περιφερειακής προστασίας. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά. Αν κανείς γνωρίζει τίποτε παραπάνω, για την αποτίμησή τους θα ήθελα να το ακούσω. Δεύτερον, για τον Ήγηρα μαθαίνουμε πολλά για τον Ήγηρα αλλά θέλουμε λεπτομέρειες ως προς την ε, που θα έχει αυτό το μελλοντικό κέντρο για προστασία, πληροφόρηση κλπ και τις εθελοντικές επιστροφές. Και τέλος, για τις επιστροφές πάλι των μεταναστών, στο Κοινοβούλιο ήμασταν αρκετά επικριτικοί για την ιδέα αυτή, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία συνυπευθυνότητα αλλά μια αρκετά ασαφής και ασυνεπής πολιτική. Ευχαριστούμε. Τέλος Μαρλίν Μπέντζη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα οι παρουσιάσεις. μπορούσαμε να πούμε τόσα πολλά πράγματα, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο θα περιοριστώ σε ορισμένα. Ιδιαίτερα τις τρεις προκλήσεις που ανέφερε ο Στρίνγκ. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο, μια τέταρτη πρόκληση επικρίνω, αντίθετα επενώ όλες τις λύσεις που προτάθηκαν για τη διάσωση ζωών, για την χορήγηση ενός αληθινού μέλλοντος στους πρόσφυγες και μετανάστες, ακόμη και τις στρατιωτικές λύσεις τις δέχομαι, αλλά χάσαμε, ξεχάσαμε το τέταρτο πρόβλημα, αυτό που έχουν στις χώρες τους οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχει εδώ μαγική λύση. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν σύραξη πρέπει να έχουν άλλη μεταχείριση από, εκείνου από εκείνους τους που φεύγουν για οικονομικούς λόγους. Τι κάνουμε για να έχουν ένα μέλλον αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες τους. Ξέρουμε αν τα χρήματα που δίνουμε επενδύονται και αν ωφελούνται οι κάτοικοι. Γιατί αν θέλουμε μέλλον στη χώρα τους να έχουν οι άνθρωποι αυτοί, μόνο τότε θα το λύσουμε. Και η μετανάστευση είναι σύμπτωμα και όχι λόγος. Γιατί αν υπάρχει πλημμύρα μπορεί να δώσουμε σφουγγάρια και σκούπες και οτιδήποτε στον κόσμο αλλά το καλύτερο θα ήταν να δούμε από πού προέρχεται η διαρροή ποιος είναι ο λόγος της πλημμύρας Άρα είναι σύμπτωμα και όχι λόγος η μεταναστευτική έξοδος. Πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα να το λύνουμε, όχι αύριο. Ευχαριστώ. Αν το είχαμε κάνει πριν από 10 χρόνια δεν θα τα λέγαμε σήμερα αυτά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την υπομονή τους και τις ερωτήσεις τους. Οι τρεις ομιλητές τώρα ας μην απαντήσουν αν δεν θέλουν σε κάθε μία από τις απαντήσεις γιατί θα γίνουν και άλλες ανταλλαγές. Ο σκοπός είναι να ωφεληθούν οι εισηγητές. Υπήρχαν όμως και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που αυτά θα έπρεπε να απαντηθούν κάθε αυτά. Είδα ότι παίρνατε τις σημειώσεις, άρα παρακαλώ ε, περιοριστείτε στα σημαντικότερα. Έχουμε μέχρι τις μία. Τα συγκεκριμένα λοιπόν κυρίως να απαντήσετε. Ο κύριος Σεράνο Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να τονίσω, όπως είπα και στην αρχή, πως συμφωνώ απόλυτα με το ότι η ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, μετανάστευσης, ούτε με αστυνόμευση, ούτε με τίποτα άλλο. Η ανάπτυξη και η συνεργασία είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά να αναπτύξουν ε, ισχυρούς ε, θεσμούς, καλή οικονομία και όπως είπατε και αρκετοί από εσάς, προσπαθούμε να Έχουμε διάφορα προγράμματα κατάλληλα για την κάθε χώρα και επίσης προσπαθούμε να ε, γίνονται όλα αυτά με όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια, διότι η διαφάνεια φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τον ε, περιορισμένο μας προϋπολογισμό. Φυσικά, ό,τι δαπάνες γίνονται για κάποια στρατιωτική επιχείρηση και να σας πω ότι μόνο μία έχουμε ε, που σχεδιάζουμε, γίνεται ε, μέσω κοινή χρηματοδότησης από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται χρήματα να ε, αντλούνται από διάφορους ε, άλλους πόρους. Μόνο λοιπόν από το Ταμείο Αθηνά. Ας μην λοιπόν έχετε ανησυχία γι' αυτό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκτός από την στήριξη στις διάφορες οικονομικές προσπάθειες και άλλα έργα, για παράδειγμα στην Σομαλία, στην Τινησία, στο Μάλι, στην Αιθιοπία, γίνονται πάρα πολλές δράσεις έτσι ώστε να, να τονωθεί η οικονομία και να προωθηθεί η σωστή διακυβέρνηση, διότι η σωστή διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι χώρες θα προχωρήσουν. Και με χαρά μου θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά τη διπλωματία τώρα, δεν ξέρω κύριε Υπουργέ, ίσως λείπατε όταν άρχισε την παρέμβασή μου, αλλά θα επαναλάβω ότι η διπλωματία είναι το κύριο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Και θα απαντήσω σε ένα από τα σχόλια του Προέδρου σε αυτό. Σίγουρα η ύπατη εκπρόσωπος είναι μία από τις πιο δραστήριες και είναι επίσης μία από τις πιο κατάλληλες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Βρίσκεται παντού. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο υπήρχε μία διάσκεψη για συνεργασία με τις χώρες του κόλπου. Η ύπατη εκπρόσωπος ήταν εκεί. Βρίσκεται στο επίκεντρο των ε, εξελίξεων. Επίσης πιστεύω ότι από αυτά που ακούσαμε όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα είναι απλό. Όταν η Ισπανία προσπάθησε να διαχειριστεί την κρίση στα Κανάρια νησιά, ήταν καλό που απετράπει μία στρατιωτική επέμβαση. Οι προκλήσεις όμως που έχουμε ε, στα μέτωπα της Λιβύης και της Συρίας είναι τελείως διαφορετικές. Κάποιοι από εσάς επίσης ανέφεραν την ανάγκη αύξησης της ανταλλαγής πληροφοριών για τις ε, μεταναστευτικές οδούς. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Μετανάστευση ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί σε ισχύ σύντομα. Επίσης, ε, χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω πως χρειάζεται δράση. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ατζέντα που είναι μη παρεμβατική, αλλά αντίθετα ενθαρρυντική για να γίνουν οι σωστές αλλαγές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε όμως να διακόψουμε τη συνεργασία με κάποιες χώρες ε, της, Ανατολική της Ανατολικής Αφρικής, για παράδειγμα, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ε, μετανάστευση. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό το διέξοδο στη Λιβύη. Σίγουρα πρέπει να επιμείνουμε και να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις ε, αρχές. Και εδώ θα ήθελα να συγχαρώ ξανά την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας για τη δράση της. Υπάρχουν ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Εθνών. Στην Λιβύη έχουμε επαφές, αλλά ως προς το μέλλον της κατάστασης και τον μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, το πώς θα καταφέρουμε να θέσουμε σε ισχύ όλα αυτά τα προγράμματα αν δεν υπάρχει κάποια αρμόδια αρχή, κάποια επίσημη αρχή με την οποία να συνεργαστούμε. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου που αναφέρουν τι μελιγενέστε σε τέτοια περίπτωση. Όμως πρέπει να περιμένουμε να δούμε το ψήφισμα όταν αυτό παρουσιαστεί. Σχετικά τώρα με τα στάδια της ε, επιχείρησης. Θα σας παραπέμψω εδώ στην απόφαση του Συμβουλίου από τις 18 Μαΐου του 2015. Εδώ αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και θα βρείτε όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας στον ιστότοπο του Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, όμως νομίζω πως ήδη χρησιμοποίησα πολύ από το χρόνο για όλους τους προσκεκλημένους. Να σας διαβεβαιώσω όμως πως θα είμαι σε επαφή μαζί σας και διμερός για να σας δώσω οποιασδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες στις επόμενες ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνοπτική σας απάντηση. Ελπίζω να ξανάρθει εκπρόσωπος της ΙΕΔ να μας μιλήσει και άλλη φορά. Ο κύριος Λέσης Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ καλές ερωτήσεις ε, και βεβαίω θα τις σκεφτούμε όταν ξαναπάμε στη δουλειά μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω δύο-τρεις. Να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Κέγγε. Εμείς θεωρούμε πως η επαναγκατάσταση δεν πρέπει να περιορίζεται σε δύο χώρες, ε, πρέπει να βασίζεται στην ανάγκη και την αιτιολογία. Νομίζω λοιπόν πρέπει να είναι, δυνα... να είναι ευρύτερη. Το έργο Presidium επίσης που σας απασχόλησε ως Υπουργό ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί. Πρόκειται για μια επιχείρηση υποδοχής, βοήθειας ε, που κάνει η Ιταλική κυβέρνηση, ο Ερυθρός Σταυρός το Save the Children, η πατερμοστία του για τους πρόσφυγες και άλλοι ήταν στη Λαμπεντούζα και σε άλλα μέρη της Σικελίας και νομίζουμε πως ήταν επιτυχές και βοηθάει αυτούς που καταφέρνουν να περάσουν. Και θα θέλαμε ακριβώς να δούμε κάποια συνέχεια. Για το θέμα της Λιβύης είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε να ξεγράψουμε τη Λιβύη δεν φύγαμε εμεί ποτέ από την Λιβύη και μάλιστα ζητήσαμε από την Υπηρεσία Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να μας δώσει περισσότερο χώρο καθώς θέλουμε να επανέλθουμε. Το προσωπικό μας στη Λιβύη με τον επικεφαλής εκεί πέρα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Κοιτάμε, παραδείγματος χάρη διάφορα έργα. να συναντήσουμε τους δημάρχους, οι οποίοι συχνά ε, βλέπουν τα ζήματα πιο άμεσα από τους υπόλοιπους ε, πολιτικούς ε, με όλο τον σεβασμό. Για να δούμε τι γίνεται και με την διακίνηση αλλά και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σεράνο για τον Νίγηρα και το μηχανισμό του Νίγηρα. Ελπίζαμε να ξεκινήσει. Υπήρχε το μνημόνιο του Οκτωβρίου 2013 για τα κέντρα υποδοχής ε, στην Λιβύη. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να πάρει τη βάρκα για να περάσει την επεξεργασία στην Λαπεντούζα. Μπορεί να γίνει αυτό στη Λιβύη. Δηλαδή αν είναι κανείς οικονομικός μετανάστης ή αν πάει στη Σκανδιναβία να βρει την οικογένειά του όπως κάνουν πολλοί Σύριοι. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει μέχρι να επαναληφθούν αυτές οι συνομιλίες οι οποίες μόλις βεβαίως ακυρώθηκαν. Ένα άλλο ερώτημα που έλεγε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αναθέσει σε άλλον τα προβλήματα της σύμφωνο πλήρως. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό. Αυτό συμβαίνει στην Ασία όπως ξέρετε. Δεν είμαστε υπέρ η δυσκολότερη ερώτηση, την οποία δεν μπορώ να απαντήσω, είναι το τι κάνουμε για τα προβλήματα στις χώρες προέλευσης. Είναι ένα μακροπρόθεσμο ζήτημα, σχετίζεται με την ανάπτυξη, την ε, σωστή, τη χρηστή διοίκηση και άλλα ζητήματα. Δεν θέλω να ασκήσω κριτική στη Frontex, εξάλλου μίλησα εγώ στην τελευταία τους διάσκεψη στην Βαρσοβία, αλλά στις παρατηρήσεις μου μίλησα για μια ανθρωπιστική διαχείριση των συνόρων. Δεν θα αμφισβητήσω εγώ βεβαίως την εντολή τους που είναι έλεγχος των συνόρων, αλλά οπωσδήποτε όταν έχουμε κατάσταση, μια κατάσταση σαν τη σημερινή, ε, ανθρωπιστική διαχείριση είναι διάσωση. Το πρόβλημα με τη Frontex είναι πως δεν ε, υπάρχει σύγκριση με την ε, Mare Nostrum γιατί είχε ξεκινήσει με 6 πλοία ενώ η Μάρε Νόστρουμ είχε 32 ελικόπτερα και υποβρύχια και διάφορα τέτοια πράγματα οι Ισπανοί, οι Ιταλοί έδιναν 9-10 εκατομμύρια το μήνα και έλεγαν ας λειτουργήσει η Ένωση ως Ένωση και να μοιραστούμε την ευθύνη. Ε, δεν έγινε αυτό με την επιχείρηση τρίτων και ελπίζω τώρα με τη νέα μεταναστευτική ατζέντα να λάβουν αυτά τα οποία χρειάζονται για να φτάνουν και παραπέρα από 35 μίλια από τις Ιταλικές ακτές γιατί στην ανοιχτή θάλασσα χάνονται οι ζωές. Γνωρίζω, έχουμε σχέση με τη Frontex, ε, τους στηρίζουμε αλλά δεν θεωρούμε πως η επιχείρηση τρίτων τα καταφέρνει όσον αφορά τις διασώσεις και ελπίζω τώρα να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση. ποσόστοση των 20.000 ένα πρώτο καλό βήμα θυμάμαι όταν μίλησα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, είπα πως έχω καλά και κακά νέα τα καλά νέα είναι πως άκουσα πως τα 13 κράτη-μέλη είναι χώρες ε, επαναγκατάστασης αλλά ε, συνολικός αριθμός των ατόμων που επαναγκαταστάθηκαν είναι 5.000 Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό ως αφετηρία και βεβαίως με ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει κανείς για μεγαλύτερο λόγο και μπορεί να κάνει περισσότερα με τρόπο πιο ανθρωπιστικό. Νομίζω ξεπέρασα το χρόνο μου, θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης και την ε, ε, υπηρεσία σας που σήμερα την εκπροσωπήσατε και τον κύριο Μουραντίνο πρέπει να ευχαριστήσουμε. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, αλλά επειδή είναι τόσο έμπειρο, ε, νομίζω ότι μπορεί να δει το διαχείριση τόσο λίγο χρόνο. Μουραντίνος έχω κάποιε απαντήσει για τα πρωτα πρώτα-πρώτα για την Λιβύη. Όλοι ξέρουν πόσο περίπλοκη υπόθεση είναι. Εγώ όμως θα συνεβούλευα υποστήριξη του Μπρέναντο του καλού μου φίλου από τον ΟΗΕ, για τη διακυβέρνηση της χώρας. Θα πρέπει κάτι να γίνει και είναι δύσκολο. Πρώτα απ' όλα έλεγχος των συνόρων, όχι μόνο από πλευρά Μεσογείου, αλλά για όλη την περιφέρεια, για όλη την γραμμή της χώρας. Και επίσης οι όμορες χώρες μπορούν να ενισχύσουν τους ε, ελέγχους αυτούς. Δεν θα πρέπει να μπαίνει κόσμο στη Λιβύη, ούτω ώστε έτσι πιο εύκολα να μπορούν κατόπιν να περάσουν στην Ευρώπη. Δεύτερον, θα πρέπει κανεί να έρθει σε επαφή, όπω είπε ο κύριο ε, Σφίν, με αυτούς τους, τους ειδικούς, τους, τις περισσότερες πληροφορίες που ξέρουν πώς να εντοπίσουν τις μαφίες. Όλοι εμεί οι Δυτικοί θα πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε, θα πρέπει να αλλάξουμε τι μεθόδου μα για τη διπλωματία. Η διπλωματία του 21ου αιώνα θα είναι η διπλωματία του ρίσκου, του κινδύνου. Γιατί να είναι κανεί ε, παρόν εκεί θα είναι επικίνδυνο, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει, να είναι σίγουρο ότι θα είναι εκεί για να λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να είναι εκεί επιτόπου τόσο ώστε να μπορέσει να αποσπάσει εκεί επιτόπου κάποια αποτελέσματα. Δεύτερον, οι αιτίες, όπως είπε η κυρία Κέλλερ, μας είπε για την πολιτική μας προς την Αφρική. Μεσοπρόθεσμα, προπόνηση πολιτική, εντάξει, αλλά θα πρέπει κάπως να αρχίσουμε, γιατί δεν είπαμε. Θα πρέπει να κάτσουμε να αναφερήσουμε όλα τα σχετικά με τη συνεργασία, το εμπόριο με την Αφρική, να, να ξεκινήσουμε μια λευκή σελίδα γεωργικές συμφωνίες, ελευθερικές συμφωνίες, ε, συμφωνίες ελευθερού εμπορίου. Όλα αυτά να τα προσαρμόσουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μια καινούργια σχέση με τις χώρες της Αφρικής. Και αυτό θα είναι το μέλλον των σχέσεων μας. Ευρώπη, Μεσόγειος, Αφρική. Κάθετη δομή και το συντομότερο, το καλύτερο. Συμφωνώ επίσης με την κυρία Πιόρκα. Για μένα ήταν η πιο μεγάλη έκπληξη ότι δηλαδή δεν είδα να υπάρχει κανένας είδου ε, μέρημνα για την πολιτική επίλυση των ε, συγκρούσεων και Ξέρω ότι κάνει πάρα πολλά, είπατε εκπρόσωπο. και την υποστηρίζω 100% στα όσα προσπαθεί. Αλλά επί τέσσερα χρόνια ήμασταν ε, απόντε από την Μέση Ανατολή. Άρα ήρθε η ώρα να κινηθούμε. Άρα να πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Τέλος. Κύριε Γκίον, μας είπατε για τη συμφωνία αυτή που αφορά τον επαναπατρισμό ή επανεισδοχή. Θα θυμάστε, είχαμε μια τέτοια συμφωνία στην Ισπανία για την επανεισδοχή. Και έτσι έγινε μια στροφή προς ε, συμφωνίες νέας γενιάς με τις ε, διάφορες χώρες. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θεωρήσει όλες αυτές τις συνθήκες και συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης και ε, διέλευσης διαμετακόμισης. Τέλος δε, θα πρέπει να συμφωνήσω με τον Πέδρο Σεράνο Χρειάζεται μια συλλογική, σφαιρική, ολοκληρωτική, ολιστική που λένε στα αγγλικά προσέγγιση. ευχαριστώ πολύ.